necessity to allow people to cover their basic living costs before you started seizing assets and so forth uh, was a socialist amendment from, uh, that I accepted. Είναι κάτι το οποίο δέχθηκα μετά από επαφή με την ΠΕΡΕΣ. Ίσως αυτό να είναι κανόνα σε ορισμένες χώρες όπως τη Γαλλία. Δέχτηκα λοιπόν αυτά τα οποία είχε πει ο κύριος Στόλογιαν αν και υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ε, εδώ παρεμηνίας, Πάντως πρόθεσή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πλήρης δημοσίευση όλων των στοιχείων ενός λογαριασμού, αλλά μόνο του τμήματος των στοιχείων που μπορεί να έχουν σχέση με τις διεκδικήσεις ή με τους ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί. Και εννοώ διαδικαστικά και δικαστικά. Αν σαν παράδειγμα 500 ευρώ είναι κάτι το οποίο διεκδικείται αλλά είναι και το κατώτατο όριο για το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία των λογαριασμών, είναι ένα όριο δηλαδή κάτω από το οποίο δεν λειτουργεί η διαδικασία αυτή, ίσως είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να διαφοροποιηθούμε και θα ήθελα να εξηγήσω στον εισηγητή ποιες ήταν οι θέσεις τις οποίες είχαμε στην προηγούμενη, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εντολής. Οι άλλες τροπολογίες νομίζω ότι δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει μια ενιαία αγορά είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα διασυνοριακής ε, συλλογής, εν πάση περιπτώσει, των χρεών μετά από τις κατάλληλες δικαστικές και διαδικαστικές ε, ε, ε, τα στάδια στα οποία πρέπει να περάσει η διαδικασία αυτή. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτεται και το κόστος το οποίο δημιουργείται από την αναζήτηση, την ανείχνευση και την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Θα ήθελε κάποιος να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με την έκθεση Στόγιαν, ε, ε, πού βρισκόμαστε λέει ο κύριος Σμιτ. Είμαστε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Ε, είστε ο εισηγητής των φιλελευθέρων και έχετε καταθέσει τροπολογίες κύριε Σμιτ αν θυμάστε. Έτσι και αλλιώς μπορείτε να πείτε ότι συμφωνείτε με τις τροπολογίες, μην ψάχνετε. Ναι, ναι, συμφωνώ, λέει ο κ. Σμιτ. Λοιπόν, συνηθίζεται, λέει η κυρία Πρόεδρος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος που έφτασε τώρα μόλις στην αίθουσα θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Στόλογιαν για μια ακόμη φορά. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, λέει ο κ. Στόλογιαν. Συνεπώς η έκθεσή σας ολοκληρώθηκε. Ε, το σημείο 7 δηλαδή. Η ψηφοφορία θα γίνει αργότερα μετά τις 11. Περνάμε τώρα στο σημείο 8. Η τροποποίηση του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι η εξέταση σχεδίου έκθεσης. Ο κύριος Γκοζές, ευχαριστώ πρόεδρε. Βλέπω ότι σιγά σιγά έρχεται πλήθος μεγάλο για τις υπηρεσίες αξιολόγησης, για τους οργανισμούς αξιολόγησης. Θα είμαι σύντομος. Όταν έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων γύρω από την έκθεση αυτή, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές αρχές να είναι σε θέση να ασκήσουν τις εξουσίες τις οποίες έχουν στα πλαίσια του συστήματος νέου από την 1η Ιανουαρίου του 2011 το νέο σύστημα που έρχεται. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίστηκα σε ελάσσονες τροπολογίες διευκρινιστικού τύπου παραμένοντας στο κεντρικό θέμα με το οποίο ασχολείται η τροποποίηση του κανονισμού, την οργάνωση δηλαδή της λεγόμενης εποπτείας. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τις υπηρεσίες αξιολόγησης. Κάποιες πρόχειρες σκέψεις και κριτικές επίσης ακούγονται γιατί αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης έπαιξαν ένα αρνητικό ρόλο για την οικονομική και δημοσιονομική κρίση την οποία βιώνουμε. Αν είχαν ένα τέτοιο πολύ κακό ρόλο τότε θα είχαμε βρει τον αποδιοπομπαίο τράγο τον οποίο αναζητούσαμε όλοι. Υπάρχουν ε, νομίζω και άλλοι ε, εμπλεκόμενοι όπως οι θεσμικοί επενδυτές και οι οποίοι με τις συμπεριφορές τους και τις αναλύσεις τους έχουν συνεισφέρει τα μάλα στην γιγάντωση της κρίσης αυτές. Λοιπόν από αυτή την χαλάρωση των κανόνων εποφελήθηκαν οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί αυτοί και όπως είπε ο Ζαν Πιέρ ο οποίος είχε αφήσει αξέχαστες αναμνήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της γαλλικής ε, προεδρίας είπε ότι θα πρέπει οι επενδυτές να, να απαλλαγούν εν πάση περιπτώσει και να απεξαρτηθούν από τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες οργανισμούς αξιολόγησης, γιατί πολλές φορές θα λέγαμε βαθμολογούν υπερβολικά και είναι πολύ πιο δραστήριες από όσο θα έπρεπε. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να αρχίσουμε και εμείς να αξιολογούμε τις υπηρεσίες αυτές αξιολόγησης και να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε ο χρηματοπιστωτικός κόσμος να μην εξαρτάται για τις αποφάσεις τις οποίες θα λαμβάνει αποκλειστικά από τέτοιου τύπου προτάσεις. Ας προσπαθήσουμε τώρα σύντομα να αντιμετωπίσουμε το θέμα του τροποποιωτικού κανονισμού. Είχα προτείνει, αν ενθυμίστε και είχε γίνει δεκτό, να υπάρξει μια έκθεση πρωτοβουλίας για, τις, για τους οργανισμούς αξιολόγησης. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής θα μιλήσουμε και άλλα θέματα, υπηρεσίες εποπτείας, δημόσια χρέη κτλ. Και πράγματι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Αυτή η διαδικασία θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την πρωτοβουλία την οποία οφείλει να αναλάβει το 2011 για να ολοκληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις υπηρεσίες αξιολόγησης. Εγώ εξέτασα προσεκτικά και τη γνώμη της Νομικής Επιτροπής και του εισηγητή της του κ. Λέινεν. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέλφους να, να στρέψουν την προσοχή τους αποκλειστικά στο κείμενο που προβλέπει την εποπτεία και όχι να καταθέτουν τροπολογίες οι οποίες ανήκουν στην έκθεση πρωτοβουλίας την οποία θα εξετάσει το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών να είναι η 13η Οκτωβρίου, η εξέταση των τροπολογιών 26 Οκτωβρίου, επανεξέταση την 8η Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 9 Νοεμβρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αν το πετύχουμε αυτό δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα και στον τριμερή διάλογο, θα είμαστε έτοιμοι σε έφετο χρόνο και ελπίζω ότι το κείμενο θα είναι αποτελεσματικό και προς εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Αυτός είναι και ο στόχος τον οποίο όλοι πρέπει να έχουμε. Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η ευρωπαϊκή εποπτεία των αξιολογητικών οίκων είναι η πρώτη θα έλεγα αποστολή την οποία αναλαμβάνει η νέα υπηρεσία ναι. ΕΣΜΑ και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε στην αρχή αυτή ε, τις αρμοδιότητες ε, και τις εξουσίες που θα της επιτρέψουν να λειτουργήσει και να προχωρήσει την αποστολή της. Ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, συνάδελφο Γκοζές για την παρουσίαση την οποία έκανε. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κείμενο Νομίζω ότι μπορούμε ε, με, με επικοδομητικό τρόπο να συνεργαστούμε σε αυτό όπως το κάναμε και στο παρελθόν. Η έκθεση αυτή αποτελεί θα έλεγα ένα σημείο δοκιμασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεων και προτάσεων το Κοινοβούλιο θα καταστήσει θα έλεγα ζωντανή την ε, ευρωπαϊκή εποπτεία στις χρηματαγορές και θα δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να δοθεί ένας κεντρικός ρόλος στις νέες αυτές αρχές τις οποίες δημιουργήσαμε και να μην παραμείνουν κενές περιεχομένου όπως θα θέλανε πολλές κυβερνήσεις. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις με το, ε, με το Συμβούλιο έτσι ώστε να πετύχει αυτό το πακέτο για την εποπτεία και επίβλεψη είναι το πρώτο βήμα και μετά από αυτό θα ξεκινήσει ένα νέο μπραντεφέρ. Το πρώτο το κερδίσαμε. Σε αυτή τη νίκη θα πρέπει να δώσουμε δώρο θα έλεγα και άλλες νίκες από εδώ και πέρα ανατομέα. Εποφελούμε εδώ για να υπενθυμίσω ότι και στον τομέα των εισοδημάτων ορισμένες κυβερνήσεις διαδρομικά θα έλεγα προσπαθούν να κλείσουν, να ανοίξουν μάλλον ένα θέμα που έκλεισε ήδη το 2009 σύμφωνα με τον κανονισμό 2060 ε, σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες προέρχονται από τρίτες χώρες. Το σύστημα του endorsement δηλαδή το οποίο δεν έχει ακόμα καθοριστεί πλήρως θα είναι ένα αρνητικό μήνυμα και πρέπει να απορριφθεί πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχετικά τώρα με την έκθεση Γκονζές, κάποιες μικρές παρατηρήσεις. Είναι πολύ καλό το άρθρο 8, η δημοσίευση δηλαδή και πλήρης πρόσβαση στις, ε, στην, στις συμφωνίες αυτές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο ανταγωνισμού που ε, χαρακτηρίζεται ο τομέας αυτός από έλλειψη ανταγωνισμού. Σχετικά με το άρθρο 36 τώρα και τις εξαιρέσεις, θα ήθελα να προτείνω μέσα από τροπολογίες ορισμένες αλλαγές στον εισηγητή. Η επιλογή να δώσουμε την κυρωτική εξουσία στις ευρωπαϊκές αρχές της εννοώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στην υπηρεσία ΕΣΜΑ είναι κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήσεις και όχι μόνο αυτό, αποδυναμώνει την ΕΣΜΑ. Πρέπει λοιπόν εμείς να καταστήσουμε αποτελεσματική την εποπτεία μας και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε περαιτέρω κυρωτικές διαδικασίες στην υπηρεσία αυτή την ΕΣΜΑ. Σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνήθως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη και το Συμβούλιο αλλά θα πρέπει οι βασικές αρμοδιότητες ε, να ασκούνται θα έλεγα από την συγκεκριμένη νέα υπηρεσία. Δημιουργείται εδώ ένα νομικό θέμα λοιπόν. Νομίζω όμως ότι αν ορίσουμε σωστά τα, τα διακριτικά περιθώρια τα οποία έχει στη διάθεσή της η νέα αρχή θα μπορέσουμε να ορίσουμε την εμβέλεια θα έλεγα των κυρώσεων στις οποίες θα μπορεί να προχωρά. Υπάρχουν κάποιες ε, νομικές αντιρρήσεις οι οποίες λέγουν ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμως επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν νομικά τη δική μας θέση ότι η νέα υπηρεσία θα είναι αυτή η οποία θα έχει την κυρωτική αρχή. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Ζων Πολ Γκοζές που βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό διότι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι, έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα ιδίως ε, με την οδηγία των investment managers και εδώ ουσιαστικά πρόκειται για προσαρμογές τεχνικού είδους και ε, ε, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα στις αρχές του επόμενου έτους, ιδίως όσον αφορά τις εταιρείες βαθμολόγησης. Καταρχήν λοιπόν στα σχόλιά μου έχω να πω ότι θα πρέπει να είναι εφικτό να μπορέσουμε να αναθέσουμε τα έργα αυτά και την παρακολούθηση εις ε, εθνικές αρχές αν πρόκειται για τοπικές ή περιφερειακές ε, ε, εταιρείες αξιολογήσεως πιστοληπτικής ικανότητος. Επίσης θα πρέπει όλα αυτά να προσαρμοστούν εις τη γλώσσα του κλάδου και θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση υποχρέωση αναφοράς των εθνικών αρχών που θα πρέπει να εξεταθεί πολύ προσεκτικά. Συμφωνώ στα περισσότερα θέματα, αλλά έχω ορισμένα σημεία όπου θα ήθελα να κάνω και τροπολογίες. Το πρώτο αναφέρεται στην πρόταση που έχει διατυπώσει ώστε οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι δεν ε, έχουν ε, αναλάβει επισήμως ε, μία αξιολόγηση να μην δικαιολογούνται να έχουν την πληροφόρηση αλλά θα πρέπει στο 10% των περιπτώσεων να υπάρχει δωρεάν παροχή των πληροφοριών για να μπορέσουμε ε, να ε, αυξήσουμε τον ανταγωνισμό μη εξουσιοδοτημένες rating agencies να μπορέσουν επίσης να συμμετάσχουν και να υπάρξει ένα σύστημα κινήτρων και γι' αυτό εδώ ε, θα έπρεπε να αλλάξει και η οδηγία για τα ίδια κεφάλαια διότι η χρήση ε, μίας δωρεάν αξιολογήσεως θα πρέπει να περιληφθεί και να προβούμε και σε ένα σωστό ορισμό. Δεύτερον, δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται με τις ε, rating agencies οι οποίες ε, έχουν εξουσιοδοτηθεί από μια εθνική αρχή. Θα πρέπει να ξαναεξεταστούν ή απλώς εμείς θα ε, κυρώσουμε την ε, αδειοδότηση των εθνικών αρχών ή πρέπει να υπάρξει νέα αξιολόγηση και στην περίπτωση τη δεύτερη υπάρχει μία απλοποιημένη διαδικασία διότι σήμερα δεν ξέρουμε ακόμη πόσοι είναι οι πόροι δηλαδή πόσο προσωπικό θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε όντως να μπορέσουμε να υποπτέσουμε σωστά αυτές τις ε, ε, ε, ε, τις εταιρείες αξιολογήσεως της πιστοληπτικής ικανότητος διότι ξέρουμε ότι χρειάζεται ένα πολύ έμπειρο προσωπικό και γι' αυτό πιστεύω μετά από ένα χρόνο να πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό για τους πόρους, για τις δαπάνες προσωπικού και στο τέλος να δούμε ποια θα πρέπει πρέπει να είναι η σύσταση του προσωπικού αυτού. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αναφέρονται σε αυτές, ε, αυτούς τους οργανισμούς credit rating και ουσιαστικά πρέπει να δούμε αν ε, το οικονομικό σύστημα εξαρτάται από την πιστοληπτική αξιολόγηση. Είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουμε. Ε, είναι σωστό ο πάντοτε να πληρώνει αυτός ο οποίος αναθέτει την αξιολόγηση θα πρέπει να ε, πληρώνει και ο χρήστης. Πρέπει να δούμε πώς θα εντείνουμε τον ε, ανταγωνισμό και γι' αυτό πρέπει να δούμε αν πρέπει να υπάρξει μία λύση ιδρύματος, αν θα υπάρξει μία ή περισσότερες δημόσιες τέτοιες οργανώσεις πιστοληπτικής ικανότητας και χωρίς να θελήσω να να βαρύνω κανέναν θα ήθελα ο Ζων Πόλο και ο Ιταλός φίλος μας να είναι συνεισηγητές ε, ο άλλος συνήθις ε, ύποπτος ε, είμαι εγώ διότι εχθές είχα ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα με το Υπουργείο μας Οικονομικών όπου λέγεται, όπου ελέγχθη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα είδος μεταποιητικού οργανισμού. Οπότε <clears throat> πιστεύω ότι εκτός από αυτά τα οποία μας είπε ο Ζων θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε και πάλι το άρθρο 30, δηλαδή υπό ποιες προϋποθέσεις ε, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες αξιολόγησης μπορούν να ανατεθούν στις εθνικές αρχές. Καταρχήν για να, να επιτραπούν ορισμένα πράγματα, δηλαδή ένα μικρό γραφείο ο αξιολογήσεως δεν μπορεί να ελεγχθεί σε μία περιφέρεια από το Παρίσι και από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνεχής ανάθεση θα μπορεί να αρθεί ότι εδώ θα έπρεπε να προβούμε σε μία διευκρίνηση κατά τρόπον ώστε αυτή η διατύπωση να βελτιωθεί. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις ε, κυρώσεις και τα πρόστιμα, συμφωνώ για το 36α και το 36β και επίσης θα έπρεπε να ξαναεξετάσουμε την ε, ακριβή ρύθμιση της αρχής του τρίτου κράτους διότι και πάλι θα μας ενοχλήσουν αυτά τα οποία είπε ο Ζων Πολ δηλαδή τι ρύθμιση μπορεί να υπάρξει για πόσο χρονικό διάστημα ποια είναι η ισοτιμία όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε και πρέπει να δούμε επίσης τι γίνεται με τη ρύθμιση σχετικά με το άρθρο 8 δηλαδή τη διαφάνιση διαφάνεια. Καταρχήν όσον αφορά αυτό που είπε ο Βολφ σε το 10% γιατί δεν μου φαίνεται σωστό περιορίζομαι ε, τον ανταγωνισμό <clears throat> γιατί λέγεται ότι μόνο οι νέες ε, οργανώσεις αξιολόγησης ε, θα μπορούν να έχουν τα στοιχεία. Δεν μου φαίνεται σωστό. Θα θέλουμε να υπάρχει σωστός ανταγωνισμός στον κλάδο. Επίσης το πρότυπο αυτό των ευαισθήτων πληροφοριών που θα δημοσιεύονται σε, ένα περιορι... σε μια περιορισμένη χρήση ιστοσελίδας δεν μου φαίνεται ξυπνό θα... δεν πρέπει να είναι οι ελάχιστες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς πληροφορίες και θέλουμε να δούμε και τι στοιχεία θέλουμε να δημοσιοποιούμε και αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε μεταξύ συναδέλφων και ελπίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν γρήγορα κατά τρόπον ώστε να, ε, να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την περαιτέρω διαδικασία διότι 1η Ιανουαρίου είναι κοντά και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστούμε 24 ε, τριμερείς διαλόγους επί του θέματος και η δικιά μας πολιτική ομάδα τουλάχιστον είναι υπέρ της νόμης να προχωρήσουμε γρήγορα. Πολύ ωραία, λοιπόν, δεν έχει ζητήσει άλλο ε, το λόγο εκτός από την υποφαινόμενη, αλλά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, οπότε θα τους δώσουμε τον λόγο σε λίγο και αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να σας πω είναι κάτι επί το οποίο μπορεί να μας διαφωτίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή το πόσο έχουν να έχουμε κατά νομιμότητα για επιβολή κυρώσεων, ε, όπως ε, είπε και ο κύριος Πιτέλα, και θα πρέπει να δούμε ποιος παίρνει την πρωτοβουλία να εγκρίνει κάτι το οποίο απόκειται στη διακριτική ευχέρεια. Και εγώ θα ήθελα επομένως να υπάρχει ανεξαρτησία της ε, αρμόδιας αυτής και να δούμε τι θα γίνει στα κράτη-μέλη και έχουμε δε το άρθρο 24 το οποίο αναφέρεται σε αυτό το θέμα που όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής που έχουν αυτοί οι οργανισμοί είναι κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον είναι αυτονόητο. γιατί προβλέπεται εδώ ένα πενθήμερο το οποίο δεν ξέρω αν επαρκεί. Γιατί έχουμε την πρωτοκόλληση, έχουμε την ενημέρωση, έχουμε διάφορες διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβεί αυτός ο οργανισμός για να προσφύγει οι οποίες δεν νομίζω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα προβλέπεται. Είναι ευκαιρίες τώρα. για την υποχρέωση παροχής κάποιων πληροφοριών. Εδώ μου φέρνει στο μυαλό ένα σχήμα καρτέλ σε σχέση με το σε ποιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και ποιοι. Δεν έχουν όλοι σε όλες. Υπάρχει υποχρέωση επομένω δημοσίευσης και εδώ έχουμε κάποια όρια σε αυτή τη ρύθμιση αν θέλουμε επομένω να είναι πραγματικά ανοιχτή αυτή η διαδικασία, αυτού του είδους το website στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση όλοι δεν είναι καλύτερη ρύθμιση. Να, τα σημεία και ίσως είναι και άλλα τα οποία πρέπει να ξαναδούμε και οπωσδήποτε θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Μήπω θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Εάν όχι, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να δευτερολογήσει ο εισηγητή. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μένει μου χαρά τι παρατηρήσει σα και νομίζω ότι έχουμε κοινό στόχο, δηλαδή ότι θα πρέπει αυτού του είδου η υποπτία για αυτού του οργανισμού αξιολόγηση είναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί και να γίνει μέχρι την ώρα του 2011. Έχουμε επομένω ε, τι τροπολογίε δεδομένε και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκο κύματο. Φυσικά και συμφωνούμε και για τα άλλα σημεία ε, για, την, για, τον ανταγωνισμό, για, το κρατικό χρέος, ε, για, το, το, το, για το ειδικό βάρος αυτής της αξιολόγησης. Όλα αυτά θα τα ασθενήσουμε και Ακριβώς όπως προείπα, συμφωνώ με τον ε, εισηγητή για την έκθεση της πρωτοβουλίας. Έχουμε τη δημοσίευση αυτού του ε, εγγράφου που, στην οποία θα προβούμε ε, αυτόν τον μήνα και θα κατεβάσουμε επίση προτάσεις για να καλύψουμε όλα αυτά τα σημεία πριν έρθει το καλοκαίρι του 2011. ό,τι μπορεί να καλύπτεται από μια δύο πρωτοβουλία προσπαθήσαμε να μην τα περιλάβουμε στο κείμενο εκείνο, διότι θα πρέπει μέχρι 1η Ιανουαρίου να έχουν ρυθμιστεί αυτά τα θέματα που δεν θίξαμε. Θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν. Και αυτό θα γίνει γιατί οι θέσεις μας είναι πολύ κοντά. Παρακαλώ να μην ταράξουμε την ισορροπία που έχουμε πετύχει με τον ισχύοντα κανονισμό. Ε, εργαστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα για να κλείσουμε το θέμα μέσα σε ένα πενθήμερο να συμφωνήσουν τα τρία θεσμικά όργανα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ταράξουμε τα νερά αυτού του κανονισμού. Είναι πολύ σημαντικό να μην ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογήσεις που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουμε ορίσει. Για δε το άρθρο 8 με χαρά μας βλέπουμε ότι η συζήτηση είναι επικοδομητική θα οδηγήσει σε βελτίωση του άρθρου τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις συμφωνώ πρόεδρε με αυτά τα οποία είπατε εδώ έχουμε κάποια θέματα σε σχέση με την υπόθεση Νερόνι και σε σχέση με τις αποφάσεις που μπορεί να λαμβάνει η Επιτροπή που δεν έχουν σχέση με διακριτική ευχέρεια. Το Συμβούλιο μελετά την περίπτωση σχεδόν αυτόματης επιβολής κυρώσεων και είπαμε ότι αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, προτιθέμετα να το συζητήσουμε αλλά άπαξ και παραμένει η διακριτική ευχαίρεια των ε, επιστολικών οργανισμών πάρα πολύ περιορισμένη. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκχωρήσουμε σημαντικές αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Όμως, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο τι αναθέτουμε και τι προβλέπουμε για την κάθε υπηρεσία, κάθε αρχή, για την ΕΣΜΑ. Είπαμε να μην έχουμε νέα αδειοδότηση έγκριση, άπαξ και έχει εγκριθεί, αναγνωριστεί κάποιος ε, οργανισμός πιστοληπτικό, πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και επίσης θα το ξαναδούμε και αυτό το θέμα όταν προχωρήσουμε σχέτω στο κειμένο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Θα ήθελα να πω στον Τζάνι Πιτέλα ότι όπως και αυτός νομίζω ότι η μάχη την οποία κερδίσαμε είναι μια μάχη που δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκύψουμε σε αυτούς που θέλουν να αποσαρθρώσουν τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να ισχύουν το 2009. Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται σήμερα και οι απορίες ε, ε τίθενται και τότε και δεν μπορέσαμε να βρούμε το 2009 ικανοποιητικές απαντήσεις και γι' αυτό δεν προχωρήσαμε σε κατάλληλες ρυθμίσεις. Νομίζω ότι η συζήτηση στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας θα επιτρέψει να βρούμε αρκετά έξυπνες λύσεις, ε, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Δεν πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα για τον Λίντς. Κλίντς. Δεν διαφέρουμε πολύ, τουλάχιστον σχετικά με τον κανονισμό αυτό. Και ο κατάλογος των σημείων προς συζήτηση δείχνει πόσο καλό είναι που χωρίσαμε αυτόν τον τροπιποιητικό κανονισμό από την έκθεση πρωτοβουλίας. Είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε κάπως ξεχωριστά. Για το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο τέθηκε, δηλαδή για οργανισμούς οι οποίοι επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν από τις εθνικές αρχές, αυτό έγινε σύμφωνα με την ενδιάμεση προσωρινή διαδικασία, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αυτό το οποίο ήθελε το Κοινοβούλιο, ούτε αυτό το οποίο μπορούσε να γίνει άμεσα δεκτό. Λοιπόν, ε, δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή με το τι θα γίνει με τους οργανισμούς που έγιναν δεκτοί ή εγκρίθηκαν από τις εθνικές αρχές. Το 2009 αυτό το οποίο μας απασχολούσε ήταν οι μεγάλες αυτές υπηρεσίες αξιολόγησης, οι οποίες είναι πολύ λίγες. Από τότε ήρθαν στην επικαιρότητα κάποιες μικρότερες υπηρεσίες αξιολόγησης εθνικού χαρακτήρα. Δεν ξεπερνούν τα σύνορά τους. Αυτές οι υπηρεσίες οι εθνικές αξιολόγησης δεν πρέπει να λειτουργήσουν σαν άλοθη για την αποδυνάμωση του ρόλου της ΕΣΜΑ. Είναι κεντρικός ο ρόλος της ΕΣΜΑ. Πρέπει να παραμείνει συνεκτική η νομοθεσία και η ποιότητα της αξιολόγησης στην Ευρώπη. Ναι, μεν μπορεί να υπάρξει κάποια θα έλεγα αναπομπή αρμοδιοτήτων προς τις εθνικές αυτές υπηρεσίες οργανισμούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε τις εξουσίες της ΕΣΜΑ, εξουσίες τις οποίες κερδίσαμε με πάρα πολύ αγώνα. Και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Είναι ψευδέστηση να νομίζει κανείς ότι μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα υπάρξει ουσιαστικός ανταγωνισμός. Δυστυχώς τα μέσα που απαιτούνται είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ακόμα και αν κάνουμε βελτιώσεις σε επίπεδο διαθεσιμότητας πιστώσεων, δεν νομίζω ότι θα αναπτύξουμε τον ανταγωνισμό γρήγορα. Για ένα απλό λόγο, οι επιχειρήσεις όπως και τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις θα στρέφονται κατά προτεραιότητα προς τις διεθνείς αυτές υπηρεσίες οργανισμούς και όχι προς ε, νέες υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν πείρα σε επίπεδο διεθνών θα έλεγα λογαριασμών υπάρχουν τέσσερις μεγάλες εταιρείες και δεν δίδονται ε, πολλές δυνατότητες στις μικρότερες υπηρεσίες οργανισμούς. Δεν ξέρω τώρα τι είναι σωστό και τι δεν είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Η σύγκληση λοιπόν των παρατηρήσεων των προλαλισσάντων δείχνει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία έτσι ώστε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει δεκτό με τις τροπολογίες του και να σεβαστούμε την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου του 2011 που είναι απαραίτητο να το κάνουμε αν δεν θέλουμε να αφήσουμε ελεύθερο χώρο σε στρεβλώσεις που θα προέλθουν από τις εθνικές συμπεριφορές. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. έχει ως εξής. Προθεσμία για τις τροπολογίες 13 Δεκάτου και πρόκειται να συζητήσουμε στις 26 Δεκάτου τις τροπολογίες. Εδώ λέει δεν έχει γίνει μετάφραση αυτό το σημείο που έχω. Εδώ έχει γίνει την 8η Νοεμβρίου που θα τα ξανασυζητήσουμε και στις 9 Δεκάτου θα ψηφίσουμε για να πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Να, το χρονοδιάγραμμά μας. Άρα 13 Οκτωβρίου για συζήτηση για προθεσμία κατάθεση των Ζούμπολ. Τι ναι. Αφού μιλούμε για την μετάφραση του κειμένου, πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, της Γραμματείας ε, και τους ε, άλλους ειδικού και όλους όσοι θα δουλέψουν ούτως ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη συζήτηση και όσοι δουλέψαν για να μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν όταν γίνουν τα πράγματα καλά να το λέμε για όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και τώρα προχωράμε πάρα πολύ καλά μια από το επόμενο θέμα μας είναι οι ψηφοφορίες που προβλέπεται να γίνουν στις 10 και μισή. Επομένως αποκτήσαμε με την ταχύτητά μας 45 λεπτά που περισσεύουν και θα κάνουμε διάλειμμα και θα ξαναμούμε στις 10.30. Οπότε πάω να βγάλω χθες το μικρόφωνο. Right. Welcome, welcome back Καλώς ορίσατε όλοι πίσω στη συνεδρίαση και παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Αυτοί οι οποίοι έχουν τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας παρακαλώ βάλτε στην σχισμή και όποιος δεν έχει την κάρτα μαζί να μου το πει τώρα. in a minute. Gunnar is, is, is right. He, ha- he's okay. Right. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Θα κάνουμε επομένω ε, την ε, ψηφορία. Κύριε Φέλ. Signora. It doesn't work. I can talk. Ο κύριος Φέιο κάτι λέει εκτός Πρόεδρος. Όχι να κάνουμε ένα, ένα τεστ, μια μικρή δοκιμή. Τώρα ψηφίζουμε. Όλοι θέλουν να ψηφίσουν ναι, τώρα ψηφίζουμε. Άνοιξε. Όχι, δεν δουλεύει. Όχι, λέει ο κύριο Φαϊό. Ναι, αλλά άμα σας να τρέχει ο χρόνος, για να το ξανακάνουμε. Εντάξει, όλοι έτοιμοι. Μπορείτε να ψηφίσετε και άλλοι δύο που δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Και έχουμε 35 από τους οποίους ψήφισαν οι 34. Για να το δούμε λέει ο κύριος Φαΐο. Τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Φαΐο και έχει ζητήσει το λόγο ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Φέιο. Τώρα που ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας θα ήθελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν σκιώδεις εισηγητές. Τους ευχαριστώ θερμότατα. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους ε, συναδέλφους. Όλοι που ήρθαν σε επαφή μαζί μου για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε όλα τα επιμέρους θέματα της έκθεσης και ευχαριστώ και τους συναδέλφους της Γραμματείας για τις προσπαθίες τους. Και τους συνεργάτες μας της πολιτικής μου ομάδας, γιατί είχαμε σκληρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Είχαμε πολιτικά ζητήματα που έπρεπε να χειριστούμε, να ρυθμίσουμε πολύ δύσκολα. Ακόμα και σήμερα το πρωί μιλήσαμε με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και για αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τους συναδέλφους του ΕΛΚ, οι οποίοι με υπεστήριξαν σε όλες μας τις συναντήσεις. τους ε, ενημέρωσα για το πώς προχωρούμε για αυτή την έκθεση και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι εάν μπορούσε το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τη συζήτηση και να ψηφίσει νωρίς θα ήταν καλύτερα. Τέλος πάντων τόσο μπορέσαμε, τόσο κάναμε και τώρα θα ψηφίσουμε. Σας υπενθυμίζω δε ότι έχουμε την ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου της οποίας προεδρεύει ο κύριος Φανερόν και ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους οπότε θα δοθεί η δυνατότητα να δώσουμε ένα πολύ δυνατό, ξεκάθαρο μήνυμα για το θέμα μας. Και το μήνυμα, ξέρετε, καμιά φορά είναι πιο σημαντικό από το περιεχόμενο. Πάντως, πάρα πολύ σωστό το ότι έχουμε ομοφωνία και αποφασιστικότητα. Πρόεδρος. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Πρώτα όλα έχουμε μια προφορική τροπολογία που αφορά την πρώτη παράγραφο. Συμφωνεί το ΕΛΚ, η ΑΛΔΕ, η Πράσινη, οι συντηρητικοί ρεφορμιστές, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, άποχες, εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο, παραγωγός 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 79, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Με προφορική τροπολογία του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόκειται για το 83. Το 82 καταπίπτει, διότι εγκρίθηκε το 81. Οπότε, εγκρίναμε το 83 με την προφορική τροπολογία και τώρα έχουμε ε, το, την, την συμβαστική Β. Με, την, ε, με αυτό το, το, το σχόλιο που αφορά μία προστίκη και την προφορική τροπολογία που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην συμβαστική Β. Που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γ. Σ. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Όλο το κείμενο χωρίς τις λέξεις και τα δύο και οι δύο και υπερβολικό πλεόνασμα, αυτές δύο φράσεις. Ε, πρώτα ψηφίζουμε χωρίς αυτές τις δύο λέξεις φράσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ποι είναι υπέρ του να έχουμε αυτές τις δύο λέξεις εκφράσεις στο κείμενο υπέρ κατά αποχές. Άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 95 περ κατά εγκρίνεται. Ήμκο 6 καλύπτεται και πάμε στο δέλτα χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο με το κείμενο χωρίς τις λέξεις στα αγγλικά particular in the euro area προσυνδυάζει ειδικά στην ευρωζώνη υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα το δεύτερο τμήμα με την φράση αυτή υπέρ κατά Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Τέλειωσε. 20-19. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Με προφορική τροπολογία. που αντικαθιστά κάποιο τμήμα το κειμένου, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ή, ε, προφορική τροπολογία. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο F, χωρίς την ψηφορία. Και εδώ το πρώτο τμήμα χωρίς τη φράση και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Χωρίς αυτή τη φράση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο δεν έχει τη φράση αυτή. Μια τριπλή προσέγγιση κλπ. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο. Πρώτο παράδειγμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός για το 9 της ΙΜΚΟ. Απορρίπτεται. Το 117 έχει αποσυρθεί. ΙΜΚΟ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 11. Καλύπτεται. Ε, συμβαστική. I. Πρώτα πρώτα χωρίς να λέει και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους υπέρ κατά εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές, εκεί εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα και τώρα έχουμε συμβιβαστική J, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται και πάμε τώρα στην 124. Με προφορική τροπολογία, μια τεχνική μεταβολή, εγκρίνεται το αρχικό κείμενο ε, του, του, του, του 14. Εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική K κάπα σε δύο τμήματα πρώτα πρώτα χωρίς να λέει ιδίω στην Ευρωζώνη χωρίς αυτή τη φράση δεύτερη με αυτήν πρώτο τμήμα δεύτερο ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Εγκρίνεται. Συμβαστική L. Έτσι δεν είναι. είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόληση 1 εγκρίνεται. 2 καλύπτεται. 3 καλύπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 καλύπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ασχόληση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 επίσης 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 καλύπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική M, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. N, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. O, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική π. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Q. Ε, έτοιμη τελευταία στιγμή για χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα χωρίς να λέει. Πώς είπατε. από εκεί που λέει ε, να συγκροτηθεί μέχρι εκεί που λέει ε, συμφωνημένος ρυθμός, ταχύτητα. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές και αυτό εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην ε, συμβαστική R, ρο. Πρώτο τμήμα. Από εκεί που λέει. Ε, να θεσπίσουν μέχρι εκεί που λέει σε επίπεδο της Ένωσης το δεύτερο τμήμα είναι ε, μετά την άνω εκεί που λέει επί προσθέτως κλπ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην συμβαστική S. Πρώτο τμήμα. Χωρίς να λέει στην Ευρωζώνη ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα στην Ευρωζώνη. αποχέ, υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στη συμβαστική ΤΑΦ. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 171. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική U. Για ποια θέλετε έλεγχο, για το 171. Ναι, έλεγχος. Διαγράφει, δεν κατέπεσε. Ψήφισαν όλοι. Ναι. U. Συμβαστική U. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 176 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει έλεγχο για την ψηφορία επί του 179. Εγκρίνεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο. 15. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 181. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183. Ως προσθήκη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 184. Απορρίπτεται. 185. Υπέρ κατά αποχές. 186. Απορρίπτεται. Προηγούμενη είχε εγκλήθει. Και τώρα έχουμε το Β συμβαστική. Το πρώτο τμήμα. Ε, η αυξάνεται μέχρι ευρωζώνη, περ κατά αποχές εγκρίνεται και μετά που λέει ειδική προσοχή μέχρι ευρωζώνη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Χ. X Έχουμε και μια προφορική τροπολογία για να απαλληφθεί η τελευταία φράση που λέει αυτός ή αυτή πρόκειται να συμμετάσχει όσον αφορά την συμμετοχή της Επιτροπής ε, στο Συμβούλιο, του ΕΚΟΦΗΝ και το Eurogroup. Ε, συμφωνεί με την προφορική τροπολογία. Ωραία. Αυτό θα είναι εκτός του τελικής ψηφορίας το, η διάταξη X εγκρίνεται. Επομένω έχουν προβλητοπολία και όχι κατά τη ψηφοφορία και τώρα έχουμε το 95 υπέρ. 195 αποχέ ε, υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, ήμικο 17 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική ύψιλον υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Για να δούμε τι λέει εδώ. Θέλει προφορική τροπολογία ή κατά διάρκεια ψηφοφορία. το πρώτο το κείμενο χωρίς τη φράση. Ε, χωρίς αναδιάρθρωση κλπ. Ποιοι θέλουν το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Μα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφορία, ούτε στο λόγο. Ε, συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή έχω κάποια σύγχυση όσον αφορά το δεύτερο μέρος. Ε, όσον αφορά το δεύτερο μέρος, μήπως μπορούμε να το επαναλάβουμε, δηλαδή στην επανάληψη της ψηφοφορίας. Μπορείτε να μου πείτε εάν ε, το συν και το πλήν αναφέρονται στη διατήρηση του κειμένου ή στη διαγραφή του κειμένου, διότι νομίζω ότι δεν ήταν σαφές στη δεύτερη ψηφοφορία για τους τους συναδέλφους για ποιο, γιατί ε, ψηφίζανε. Πρόεδρος, έτσι κι αλλιώς θα κάναμε επαλήθευση γιατί ήταν ωριακή ψηφορία. Όλα τα άλλα τα πήγαμε καλά. Λοιπόν, πρώτα πρώτα τι κάναμε. Ψηφίσαμε το κείμενο χωρίς αυτή τη φράση. Και κατόπιν ε, ψηφίσαμε για το κατά πόσο θέλουμε να υπάρχει αυτή η φράση. Και κατόπιν είπαμε συν, ε, που σημαίνει θέλετε, και αν βάλετε πλην, σημαίνει ότι δεν θα είναι αυτή η φράση μέσα. Εσείς θέλετε να μην υπάρχει αυτή η φράση, αλλά θέλετε το πλήν. Για να δούμε τώρα, θα κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί ήταν ενεργική ψηφορία. Μόνο το δεύτερο τμήμα για το πρώτο τμήμα το εψηφίσαμε και ενεκρίθη. Ωραία, δεν πρόεδρο. Από ό,τι βλέπουμε έχει μετακίνηση των ψηφισάντων. Τι θέλετε, θέλετε το λόγο. Ο εισηγητής. Ψηφίζουμε, Πρόεδρε, την φράση που αρχίζει εκεί που λέει On Ordinary Resolution of Sovereign Debt. Υπέρ κατά. Όμως, Πρόεδρε, από ό,τι Κατάλαβα, Πρόεδρε. Ψηφίσαμε το πρώτο και το τρίτο τμήμα στην αρχή και τώρα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Το ΕΛΚ είναι υπέρ του πρώτου τμήματος και του τρίτου και κατά του δευτέρου τμήματος. Πρόεδρος. Ναι, είπαμε. Όλο αυτό εκτός από εκεί που λέει ότι θα γίνει μία ε, έφτακτη ρύθμιση του κρατικού χρέους. Φερρυπίν αναδιάρθρωση αυτού. Orderly resolution. Συν, παναπεί, θέλετε αυτή τη φράση, πλην, χωρίς αυτή τη φράση στο κείμενο. I think that that's uh, pretty obviously that they're not in. Okay, so now we can move on to amendment 208. Τώρα πάμε στην τροπολογία 2008 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, δεύτερη τροπολογία του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το αρχικό κείμενο ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2010 υπέρ, 210 με συγχωρείτε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο συμβιβαστικής α εγκρίνεται, β εγκρίνεται. Έχουμε ΖΑ και ΖΒ. 211 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ZC ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ZD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ZE ZE ε, με μία προφορική τροπολογία των πρασίνων όπου προστίθεται ε, μετά από τη φορολογία επιχειρήσεων με εκτενείς διαδικασίες ενάντια στον αθέμητο ανταγωνισμό στα θέματα φορολογίας για να διευρυνθεί η άμεση ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Με αυτή την προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στην ε, ε, ZF χωρίς, στην αρχή χωρίς τις ε, δύο πρώτες λέξεις και στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί. Εγκρίνεται το πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πρέπει ουσιαστικά να μετράμε τα χέρια και όχι του συντονιστές ε, ΙΜΚΟ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, ZG με μία, ε, ένα διαχωρισμό της τελευταίας στιγμής. Το πρώτο χωρίς τις ε, λέξεις and assess the feasibility και το δεύτερο μέρος αυτές τις λέξεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη αλλά ας κάνουμε έναν έλεγχο. Επειδή ορισμένοι απέχουν είναι πιο συγκεχημένη εικόνα. Απερίφθη. Και τώρα προχωράμε στην 220 241. 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη αλλά δεν είμαι βέβαιη οπότε παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος όντως απερίφθη απασχόλησης 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 καλύφθηκε Παράγραφος 1, κεφάλαιο 7, ε, εγκρίνεται, συμβιβαστική ζήτα ε, γιώτα. Το αρχικό κείμενο της, ε, του παρατήματος 1 εγκρίνεται, 2.49 ε, εγκρίνεται, 250 δεν είναι αποδεκτή, άρα το κείμενο το αρχικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 251 απορρίπτεται, αρχικό κείμενο εγκρίνεται 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ σε δύο μέρη πρώτο μέρος χωρίς ε, το κείμενο «And developing ideas for the reform of the treaties» και δεύτερο μέρος με αυτό. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η παραπομπή στο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εκτιμώντας ένα και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 3 ε, καλύπτηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης το, η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίθηκε. Τώρα προχωράμε εις ε, ε, ε, στα εκτιμώντας 5 μέχρι 13 εγκρίθηκαν τροπολογία στο εκτιμώντας 5 εγκρίθηκε η ε, τα εκτιμώντας 15 έως 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, εκτι, η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 ε, είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά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 εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ZJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία C ε, απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ZK υπέρ κρατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ε, συμβιβαστική ZL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ZM σε δύο μέρη στο πρώτο μέρος ο, μέχρι το pursuit υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική ζεντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, ΙΜΚΟ 3 έχει καλυφθεί. Να ψηφίσουμε τώρα το αρχικό κείμενο. Ωραία. Για το εκτιμώντας I. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική ε, ε, ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ένα αύκο εσύ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αύκο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 65, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ZP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ZQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο γνωμοδότησης. Προσθέτει αυτές τις λέξεις στο τέλος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, το γνωμοδότηση της Επιτροπής Προπολισμού Α ε, καλύφθηκε. Ε, για να δούμε την β προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται C ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική προφορική τροπολογία του εισηγητή που συμφωνούν όλες οι ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα στο κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. ...32 υπέρ, 6 κατά και 3 αποχές. Συγχαίρουμε τον κύριο Φέγιο. Καλώς περνάμε στο σημείο 10 παρακαλώ. Έχουμε τώρα την ψηφοφορία για την για γνωμοδότηση του κυρίου Στόλογιαν. Θέλετε να γίνει ομαδική ψηφοφορία των τροπολογιών. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, λέει η Πρόεδρος. Γιατί υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τροπολογία 4 Λοιπόν, παράγραφος 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 4. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, δεκτή. Παράγραφος 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογημένο το κείμενο. Ηλεκτρονικά παρακαλώ θα ψηφίσουμε την τροπολογημένη γνωμοδότηση Στόλογιαν. 41 υπέρ. Απόλυτη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια και Στόλογιάν. Καλώς. Αυτά τελειώσαμε σήμερα, το πρωί τουλάχιστον. Α, για μια στιγμή κάτι ξέχασα. Ξέχασα κάτι. Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης σε σφαιρικό ευρωπαϊκό επίπεδο η κυρία Ποδηματά. Όσοι θέλουν να φύγουν παρακαλώ να το κάνουν ε, σιωπηλά. Δίνω το λόγο στην Άννη. Thank you, Sharon. Shall I start? Yes. Ευχαριστώ Σάρων. Ξεκινάω. Παρακαλώ ότι κουβέντες έχετε να κάνετε να τις κάνετε έξω έτσι ώστε να μπορέσει η κυρία Ποδηματά να συνεχίσει. Η, συζήτηση που διεξάγεται σήμερα σχετικά με τα νέα καινοτόμα... Όλα, you've got a problem. Yeah, that's Okay, Annie. Thank you. Η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για τα νέα καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης είναι μια συζήτηση που διεξάγεται όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει έρθει ασφαλώς ξανά στο προσκήνιο εξαιτίας της κρίσης, η οποία ανέδειξε τα όρια των παραδοσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων και την ανάγκη βεβαίως για νέες πηγές χρηματοδότησης. Για δύο κυρίως λόγους πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέους πόρους για τη χρηματοδότηση μεγάλων κοινών δράσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι οι στόχοι της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η χρηματοδότηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, αλλά όταν μιλάμε για την Ευρώπη ε, μιλάμε και για την ε, χρηματοδότηση των προκλήσεων που καταγράφονται στην ε, Ατζέντα 2020. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιατίας που ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο και με τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η μία πτυχή και η άλλη εξίσου σημαντική πτυχή που φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι η ανάγκη να απαντήσουμε στο αίτημα των πολιτών ε, και ειδικά των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δικαιότερη κατανομή του βάρους της ανάκαμψης και για ανάληψη μέρους της ευθύνης, μέρους του βάρους της σημερινής κρίσης από τους φορείς και τους τομείς εκείνους που φέρουν και βασική ευθύνη για την σημερινή κατάσταση. Ε, υπάρχουν ωστόσο, ε, αγαπητές συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι, δύο ακόμη σημαντικές παράμετροι ε, στους οποίους πιστεύω ότι εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη σημασία. Η πρώτη πτυχή αφορά ε, το γεγονός ότι η συζήτηση για τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία συνδέεται άρρηκτα με την πρόσφατη απόφασή μας να δημιουργήσουμε ένα νέο φιλόδοξο πλαίσιο χρηματοδοτικής εποπτείας και λειτουργίας των αγορών με βασικό στόχο την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και την επανεβεβαίωση ότι ο βασικός ρόλος, η βασική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ε, η χρηματοδότηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας. Και η δεύτερη τυχή που επίσης συνδέεται με τη συζήτησή μας για τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία αφορά την, και πρέπει να αφορά κατά τη γνώμη μου την ενεξελίξη συζήτηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει ε, να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Δύο λόγια ήθελα να σας πω ε, για το ιστορικό του πράγματος. Η έκθεση που ετοιμάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασίζεται σε ένα κείμενο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά ε, στον τομέα των νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ε, τα οποία επιμερίζει σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στα εργαλεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και μέσα σε αυτά είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο φόρος επί των, ε, επί, της, επί των χρηματοστοπικών δράσεων, το Financial Activity Tax, και ε, η μεγάλη συζήτηση για τη συνεισφορά των τραπεζών, το Bank Levi. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία αφορά ε, τη χρηματοδότηση των στόχων ε, της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και εκεί στο επίκεντρο είναι η συζήτηση για τη θέσπιση ενός φόρου άνθρακα και η τρίτη κατηγορία η αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών καινοτόμων εργαλείων ε, για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών στόχων. Ήθελα να θυμίσω, ε, εφόσον ξεκινάμε σήμερα αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή μας, ότι με βάση το ψήφισμα που έχει οθετήσει το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο, πριν από ένα περίπου χρόνο ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει και να υποβάλει μια μελέτη επιπτώσεων ε, γύρω από τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αυτή η μελέτη δεν έχει ε, ακόμα υποβληθεί. Ε, τα νεότερα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ζήτησε επίσης συγκεκριμένη ανάλυση των διαφορετικών επιλογών για την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και μέσα στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, η Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της. Σε επίπεδο Συμβουλίου γνωρίζετε ασφαλώς ότι η Βελγική Προεδρία έχει θέσει το θέμα μεταξύ των βασικών της προτεραιοτήτων, ε, γεγονός που έχει κάνει ε, σε μεγάλο βαθμό πράξη, φέρνοντας το θέμα της θέσπισης φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και της συνεισφοράς των τραπεζών στην ατζέντα των συζητήσεων σε δύο διαδοχικά ε, Συμβούλια Υπουργών Οικονομικών, σε δύο διαδοχικά Συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ. Ε, ένα ζήτημα λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, αφορά τις κατηγορίες των διαφορετικών ε, καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ένα άλλο ζήτημα που είναι ανεξάρτητο ως ένα βαθμό από την επιλογή και τις προτεραιότητες που θα θεσπίσουμε αφορά τη διαχείριση ε, των εσόδων, τη διαχείριση των πόρων που θα προκύψουν από αυτά τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, ήθελα να μείνω ε, ε, λίγο στην, στον πρώτο πυλώνα που αφορά στα εργαλεία του χρηματοπιστωτικού τομέα με δεδομένο ότι θα έχουμε μία γνώμη που θα υποβληθεί από την Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα επικεντρωθεί στα ζητήματα που αφορούν τη θέσπιση ε, του φόρου του άνθρακα ε, και επίσης θα έχουμε ε, μία γνώμη από την Επιτροπή Ανάπτυξης σε ενισχυμένη συνεργασία με την δική μας Επιτροπή για τα θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών στόχων. Σε ό,τι αφορά την, τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θέλω να μείνω γιατί είναι το ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων όλες αυτές τις μέρες και στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Ε, και να ανοίξουμε ε, τη συζήτηση και να πάρω τις θέσεις και τις απόψεις και τις αντιδράσεις σας στα ζητήματα αυτά που αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ε, ξεκινάμε νομίζω με μια γενική παραδοχή ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας σήμερα έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση σε ό,τι αφορά τη φορολόγησή του. Μεταχείριση η οποία κιόλα δεν δικαιολογείται εάν αναλογιστούμε και την, την ευθύνη του, τη συμβολή του στην πρόσφατη κρίση, αλλά και την εξίσου σημαντική στήριξη ε, που, έλαβε, που έλαβε πρόσφατα ε, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, από εθνικά κονδύλια. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποτελεί καταρχήν μια ευκαιρία, μια βάση για να αναστρέψουμε αυτό το αίσθημα αδικίας των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην ε, αντιμετώπιση, στον περιορισμό επικίνδυνων συστημικά συναλλαγών, όπως είναι οι ακάλυπτες πωλήσει, όπως είναι το εμπόριο υψηλής ταχύτητας, το high frequency trade, και ως εκ τούτου να συμβάλλει ε, αποφασιστικά στην αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αγοράς και με αυτή την έννοια έλεγα πριν ότι πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή συνδέεται άρρηκτα με τις πρόσφατες αποφάσεις μας για τη δημιουργία ε, του νέου πλαισίου εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεύτερο θέμα, ε, δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση ότι είναι ασφαλώς προτιμότερο και ευκταίο να καταφέρουμε να πετύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία στο πλαίσιο του G20 για τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η συζήτηση ωστόσο που έχει ανοίξει και η οποία ζητάει απαντήσεις από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, είναι ε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο δεν πετυχαίνουμε διεθνή συμφωνία. Ε, και αυτό ε, γιατί το να προχωράμε πιστεύω σε διαγγέλματα και σε δηλώσεις υπέρ της παγκόσμιας δράσης δεν έχει νόημα, δεν έχει αποτέλεσμα όταν δεν είμαστε ταυτοχρόνως έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει ασφαλώς πληθώρα τεχνικών ζητημάτων που την συνοδεύουν και που ζητούν απαντήσεις. Ε, ορισμένα από τα ερωτήματα που έρχονται, έχουν έρθει στο προσκήνιο αφορούν για παράδειγμα την πιθανή επιβάρυνση στην ανταγωνιστικότητα του ε, ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ε, εδώ τεκμηριωμένες απαντήσεις ε, από αρμόδια Ινστιτούτα αναφέρουν ότι ε, με έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φορολόγησης και μια καλά οργανωμένη αγορά που δίνει κίνητρα ε, στον επενδυτή να επιλέξει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης αγοράς απαντά στο πρόβλημα, στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Ένα δεύτερο, ένα δεύτερο θέμα που έρχεται στο προσκήνιο αφορά στη γεωγραφική ανισορροπία ενός τέτοιου φόρου με δεδομένο ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, είναι συγκεντρωμένες σε ένα περιορισμένο αριθμό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και εδώ νομίζω ότι μία απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι ε, επιλέγοντας να κατανείμουμε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων που θα προκύψουν από τη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου ε, στα ίδια τα κράτη-μέλη που θα έχουν και την ε, βασική ε, επιβάρυνση δίνουμε απάντηση και στο ζήτημα της γεωγραφικής ανισορροπίας. υπάρχουν και άλλα πολλά ερωτήματα που αφορούν κυρίως τεχνητές πλευρές της θέσπισης ενός φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, νομίζω ότι η συζήτηση τώρα ξεκινάει και πολλά από αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνάρτηση με τις προτάσεις που θα παρουσιάσει η Επιτροπή. Θέλω ωστόσο να επισημάνω ε, ότι ε, δεν θα πρέπει να χαθούμε στα καθαρά τεχνικά ζητήματα τα οποία ασφαλώς δεν πρέπει να υποτιμήσουμε, όπως είπα και πριν, αλλά ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ουσία και να κρυφτούμε πίσω από τεχνικά προβλήματα κατά κάποιο τρόπο ως πρόσχημα πίσω από το οποίο συγκαλύπτεται η έλλειψη ε, πολιτικής βούλησης για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ε, δύο άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη φορολόγηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τον τελευταίο καιρό, τα γνωρίζετε, ε, είναι ο φόρος της χρηματοπιστωτικής δράσης, Financial Activity Tax και, το, τα Bank Levice. Ε, ήθελα απλώ να θυμίσω ότι υπάρχει μια βασική, μια ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα σε αυτού του δύο φόρου και τον φόρο ε, επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το γεγονό ότι κατευθύνονται κυρίω και οι δύο αυτέ επιλογέ και οι δύο αυτοί φόροι προ τη φορολόγηση των κερδών και άρα εξ αντικειμένου δεν μπορούν να έχουν συμβολή, δεν μπορούν να παίξουν τον ρυθμιστικό και σταθεροποιητικό ρόλο προς τις αγορές που μπορεί να παίξει ένας φόρος επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Άρα είναι θέμα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων μας, ε, κατά τη γνώμη μου. Εάν δηλαδή θα δώσουμε το βάρος ε, μόνο και μόνο στην, στην συγκέντρωση εσόδων ή θα συνδυάσουμε το στόχο τη συγκέντρωση εσόδων με την, με την προώθηση νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων με έναν τρόπο που θα επιτρέψει παράλληλα μια ασφαλέστερη ε, λειτουργία των αγορών και ένα περιορισμό των ε, κερδοσκοπικών συναλλαγών που δεν έχουν απολύτως καμία συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Σε μισό λεπτό, Σάρων, τελείωσα. Ήθελα για το φόρο άνθρακα να πω μόνο μία κουβέντα. Ε, ένα σημαντικό τομέα των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας σήμερα φορολογούνται ακριβώς ε, με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως της ε, ενεργοβόρας ή της περιβαλλοντικά επιβλαβούς ε, λειτουργίας τους και αυτή η ουδετερότητα πιστεύω ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με, την, με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα αλλά και συνιστά μία μορφή φορολογικής αδικίας όταν άλλοι τομείς όπως αυτός της αγοράς εργασίας καλούνται να αναλάβουν σημαντικό μέρος του φορολογικού άχθους. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να επιβάλλουμε στην πράξη την αρχή ορυπαίνων με την ευρία έννοια του όρου πληρώνει, μεταφέροντας έτσι το φορολογικό βάρος από την απασχόληση στην περιβαλλοντική εμπροκειμένο μόλυνση, μέσα από την εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα σε τομείς για τους οποίους δεν έχει ισχύ, δεν έχει εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων και ε, μέσα από την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας με στόχο ε, να συμπεριληφθεί και το βασικό κριτήριο της ενεργειακής κατανάλωσης στα κριτήρια. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των στόχων της ε, ανάπτυξης, όπως σας έλεγα και πριν, θα έχουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης, ενισχυμένη αρμοδιότητα με μας ε, οπότε, στην διάρκεια της επόμενης συζήτησής μας, όταν θα συζητήσουμε και το σχέδιο έκθεσης, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιοι ομιλητές, αλλά θα δώσω πρώτο τον λόγο στους σκιώδεις. Σμιτ, Λάμπερτς και μετά θα περάσω στους υπολείπους το λόγο. Όλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για, για την πρόταση εργασίας. Στην ουσία ξεκινάμε εκ νέου μια καινούργια παρόλα αυτά συζήτηση. Είναι περίπλοκη η υπόθεση αυτή και παρουσιάζει δυσκολίες. Καινοτόμο «Τόμες χρηματοδοτήσεις είναι μια φράση η οποία προκαλεί μερικές φορές κάποιες υποψίες. Και ομολογώ ότι και εμένα δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Αλλά ταυτόχρονα το περιεχόμενο της πρότασης αυτής είναι πολλαπλό. Εμείς θέλουμε ένα σαφές σταθερό κείμενο σαν βάση. Αν αυτό είναι αυτό που επιθυμούμε, τότε θεωρούμε και μία απαραίτητη μία σταθερή ε, βάση φορολογίας. Σε αυτή την περίπτωση ξεχνάμε τη φορολογία του άνθρακα γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερα επιμέρους και λεπτομεριακό. Έχει θετικά στοιχεία βέβαια. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι το πρόγραμμα για την ανταλλαγή ποσοτήτων διοξοδίου άνθρακα δεν, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ίσως να δημιούργησε κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά παρόλα αυτά η αρχή Λειτουργία αυτού του συστήματο είναι μια καλή ιδέα. Όταν πετάω στις Βρυξέλλε, ας πούμε νιώθω ότι κάτι γίνεται πέρα από αυτό, έχει κάτι το θετικό. Τι είδου φορολογία θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε μια φορολογία η οποία να υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό θέλουμε. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μια σταθερή, μια εδρεωμένη φορολογική βάση. Νομίζω λοιπόν ότι οι χώρες και οι εκπρόσωποι των χωρών ή τουλάχιστον όσοι εκπροσωπούνται εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν στις κυβερνήσεις τους και στα κοινοβούλια τους και να τους πούμε κοιτάξτε μην αγνοείτε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχετε αναλάβει προς ε, την Ατζέντα 2020 προς τα Ηνωμένα Έθνη Βρισκόμαστε στο 0,4% στα ODA. Συνεπώς είναι πολύ λίγες οι χώρε οι οποίες ε, έχουν πετύχει το 0,7% στο οποίο έχουν δεσμευτεί. Συνεπώς είμαστε χαμηλά ακόμα. Αν οι χώρε εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους και τις συμφωνίες τις οποίες έχουν κάνει στα πλαίσια του ODA, ίσως ακούγεται περίεργα να μιλάμε για φόρους πάλι. Γιατί τους φόρους ποιος τους πληρώνει. Τους πληρώνει ο καταναλωτής, τους πληρώνει ο πολίτης τους φόρους. Δεν είναι δωρεάν η συλλογή των φόρων. Κάποιος πληρώνει από πίσω. Είμαι λοιπόν επιφυλακτικός σε σχέση με κάποιες από αυτές τις αρχές. Σχετικά με το φόρο ο οποίος προκαλεί πάρα πολλές συζητήσεις. Αν κατάλαβα αυτά τα οποία άκουσα, είπατε ότι δεν θα πρέπει εμείς να καταβληθούμε από τεχνητά προβλήματα και από την έλλειψη ε, της πολιτικής βούλησης. Δεν νομίζω ότι ε, θα δεσμευτεί κανείς από τέτοιου είδους προβλήματα. Φυσικά και είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και τις αντίθετες απόψεις κάποιοι που θεωρούν τέτοιου είδους φορολογικές επιβολές απαράδεκτες. Σαν παράδειγμα ο κύριος είπε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πιο μαζικά από όσο περιμέναμε και υπάρχουν ε, πολλές επιφυλάξεις. Πρέπει να ακούμε και την αντίθετη απόψη λοιπόν, όχι μόνο αυτοί που είναι υπέρ, πρέπει να ακούγονται αλλά αυτοί που είναι και κατά. Εδώ τώρα να πω κάτι στην κυρία Μπερές. Στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κλίντζι όπως θέλετε πείτε την, και υποτίθεται ότι εκφράστηκαν απόψεις υπέρ αυτού του φόρου για τις ε, συναλλαγές, ε, τις χρηματοπιστωτικές, τραπεζικές κτλ. Και πολλοί, ακόμα και φιλελεύθεροι, υπερψήφισαν ουσιαστικά την άποψη αυτή. Αλλά στο τέλος αυτής της συζήτησης και του κειμένου στο οποίο οδήγησε είπαμε ότι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια μελέτη επιπτώσεων και όταν αυτή η μελέτη ολοκληρωθεί τότε θα συμπληρώσουμε την πρόταση και μάλιστα σε σφαιρικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο την τελευταία στιγμή το προσέθεσαν οι πράσινοι. Είναι κάτι για το οποίο εγώ διευκολύνομαι να το υπερψηφίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να μάθω όμως ε, αν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θεωρούν ότι θα πρέπει εμείς να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ότι μπορούμε να εισάγουμε αυτόν τον νέο φόρο, χωρίς να ακούσουμε τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να περιμένουμε την άποψη της ομάδας των 20, του G20 σαν παράδειγμα. Και αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε οφείλω να πω ότι είμαι επιφυλακτικός. Πάντως, ακόμα και αυτό το οποίο αποδεχθήκαμε στα πλαίσια της Επιτροπής Κρίσης, είναι ένας φόρος ο οποίος παρουσιάζει δυσκολίες. Προσωπικά έχω επιφυλάξεις, αλλά παρόλα αυτά ε, εκφράζοντας τη φιλελεύθερη ομάδα ξεπερνάω τις επιφυλάξεις μου και εν μέρη συμφωνούμε. Σχετικά τώρα με τα bank levies, τα τέλη τα τραπεζικά, που νομίζω ότι οι συζητήσεις τώρα ξεκινάνε. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, διαφορετικά επίπεδα ε, φόρων, τελών, κυρώσεων, προστήμων, όπως θέλετε πείτε τα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε συνολικά τι θα πληρώσει ο καταναλωτής. Όλα αυτά μαζί πόσο θα κοστίσουν στον καταναλωτή. Είναι ψευδέστηση να πηγαίνει κανείς ότι θα χρηματοδοτηθεί ένα ειδικό ταμείο για αυτό το πράγμα, ένα άλλο ειδικό ταμείο για την επίλυση των διαφορών, ένα ειδικό ταμείο για την κάλυψη της ασφάλειας των επενδύσεων Εντάξει, όλα αυτά ποιο θα τα πληρώσει, ποιο θα καλύψει το κόστος. Ο πολίτη, ο καταναλωτή, ο πελάτη της Τράπεζα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αποδηματά γιατί ξεκινάει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ένα κείμενο εργασίας επαναλαμβάνω. Είπα ότι στην ομάδα μας έχουμε κάποια θέματα προς συζήτηση και προς διευκρίνηση. Κάποιοι από εμά είμαστε υπέρ, δεν θα δω τα ονόματα, θα τους αποκαλύψετε φαντάζομαι μόνοι σας. Και κάποιοι άλλοι είναι κατά, αλλά κατά. Νομίζω λοιπόν ότι ε, τις ίδιες τάσεις θα συναντήσετε και σε άλλες πολιτικές ομάδες. Θέλω να είμαι ειλικρινής, θέλω να στηρίξει ε, η πρότασή μου με ισχυρό τρόπο την πρότασή σας, η ομάδα μου την πρότασή σας. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε όμως. Dobrý den. Tak to bylo vtipné Πάρα πολύ ε, καλή χειρονομία από τον ε, μου αξιότιμο συνάδελφο Όλε Σμιτ. Πάρα πολύ ευγενικά τόσα είπε και μας είπε ότι όχι μόνο υπάρχει διάσταση απόψεων αλλά θα προσπαθήσει παρόλα αυτά να συγκεντρώσει και να εξεύρει μια συνένεση. Όλα αυτά τα οποία συζητούμε τώρα, κατά τη γνώμη μου, δείχνουν ότι η σημασία δεν έγκυται μόνο στο κείμενο κάθε αυτό, το γράμμα, αλλά κυρίως το πνεύμα του κειμένου αυτού και πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας το κείμενο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Και το αυτό που με εντυπωσίασε όταν πρωτοδιάβασα το έγγραφο ήταν το ότι χρειαζόμαστε καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης. Ο, ο είπε ότι του φάνηκαν όλα αυτά ύποπτα ναι, και σύμφωνα μαζί του, διότι όπως περιγράφεται εδώ, η καινοτόμη μορφή της χρηματοδότησης μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι πρόκειται ή για τρόπο φοροαποφυγής ή για τρόπο εξέβρεσης, επινόησης νέων μορφών φορολογίας. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε αφού υπάρχει ο τρόπος στην, στην οικονομική επιστήμη να βρούμε ένα άλλο όνομα για αυτά τα μέσα. Και επίσης, ακριβώς λόγω της ε, κρίσης, καταβάλλεται προσπάθεια εξέβρεσης νέων μορφών φορολογίας. Θα δοθεί σκληρή μάχη για τον προϋπολογισμό, ξέρετε, ή στο Συμβούλιο και είναι σαφές ότι υπάρχει ένα μπλοκ κρατών στο Συμβούλιο που διστροπούν όσον αφορά κάποιες δαπάνες που πρέπει να γίνουν. Επομένως, βλέπετε ακόμη ένα, ένα κίνητρο για να προσφύγουμε προς αυτές τις νέες μορφές χρηματοδότησης. Από την άλλη μεριά, η μεγάλη φιλοδοξία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ε, όμω δεν έχουν τα χρήματα τα οποία του χρειάζονται για να ασκήσουν τι πολιτικέ που θέλουν. Δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα από παραδοσιακέ ε, ε, πηγές φορολογία. Άρα χρειάζεται η εξέβρεση τέτοιων ε, μέσων χρηματοδότηση για να έχουμε τα χρήματα να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Κάτι άλλο το οποίο το ανέφερε η εισηγήτρια πολύ σωστά, ότι εδώ έχουμε την προσπάθεια να τιμωρηθούν κάποιοι διότι συνέβαλαν στην ε, γέννηση αυτής της κρίση. Αυτό λέει το τέλος που θέλουμε να βάλουμε στι τράπεζε. Θέλουμε να το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι φταίνε και οι τράπεζε για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Εγώ όμω δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Και παρόλα αυτά σέβομαι το ότι πρόκειται για την κυρίαρχη άποψη στην Επιτροπή μας αλλά και στο Κοινοβούλιο. Και βλέπω τρεις λόγους που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο να είναι υπέρ αυτών των καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης. Γιατί δεν αρχίζουν τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα να εξοικονομούν κάποια χρήματα. Γιατί δεν συρρυκνώνται τον προπολογισμό γιατί δεν το γράφει αυτό το κείμενο, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη με περικοπέ στου εθνικού προπολογισμού. Είδαμε τι γίνεται στα επιμέρου κρατη κράτη-μέλη. Εμείς λοιπόν εδώ είναι να το να ανήπτουμε τα σχήρα μα και να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε καμία σχέση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να, σφίγγει το ζωνάρι. Υπάρχει περιθώριο. Περικοπές σε κάποια προγράμματα, κλείσιμο κάποιων ε, υπηρεσιών που δεν χρειάζονται και μην με παρεξηγείτε. Δεν θέλω να προκαλέσω, αλλά πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσον πραγματικά χρειάζεται δύο ή τρει έδρε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πώ να εξοικονομηθούν χρήματα. Θα πρέπει ε, τα θεσμικά όργανα να κοστίζουν λιγότερο. Και να πώ θα υπάρχει λιγότερη πίεση για επιβολή νέων μορφών φορολογίας. Δεν θα τρώω να μπω στις ε, λεπτομέρειες, στην ουσία του ζήτηματο σε σχέση με τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Πάντως ξέρω ότι πάρα πολλοί ειδικοί πρεσβεύουν ότι αυτή η βάρυνση των ε, συναλλαγών πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα και να μην τα λύσει. Το θέμα θα είναι πολύ πιο μπερδεμένο από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. τον επιβαρύνουμε τις συναλλαγές είναι σαν επιβάλλουμε κάποιο είδους τιμωρία στις τράπεζες. Όχι, δεν είμαι, δεν, δεν υπέρ των τραπεζών και των hedge funds, αλλά δεν πιστεύω ότι φταίνει οι τράπεζες για την ε, κρίση. Η αγορά στην κατάσταση που βρισκόταν, εκείνη συνέβαλε στην γέννηση της κρίσης. Και η οποία χτύπησε τις τράπεζες. Τώρα όσον τα ευρωομόλογα νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθεί το ΕΚΟΦΗΝ και γενικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, και αφού τοποθετηθούν θα ξέρουμε. Θα πρέπει πάντως να περιμένουμε να ακούσουμε τι πρεσβεύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. να δούμε τι γίνεται με την ε, διάρκεια ζωή των βρωμολόγων ε, και άλλα ειδικότερα ζητήματα. Υπάρχει, ε, υπάρχουν θέματα εκεί να συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε στην πολιτική μας ομάδα. Ε, τα έχουμε ήδη συζητήσει όσον αφορά τους ε, ρεφορμιστές συντηρητικούς. Δεν σας λέω τι, ποια άποψη κατήσχησε. Να δούμε. Ελπίζω τέλος πάντων να, να βρούμε ένα κείμενο το οποίο εκπροσωπεί αυτό το οποίο πιστεύει ο μέσος πολίτης. Δεν ξέρω εάν ένα κείμενο μπορεί να αντικατοπτρίζει την άποψη όλων των πλών πολιτών. Οπότε θα ξεκινήσω και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ τον όρο αυτό παρατηρώντας ότι όταν συζητάμε για οικονομική διακυβέρνηση ε, δεν έχουμε ε, επαρκή απαρτία και λυπούμε διότι το ΕΛΚ ε, δεν ε, εκπροσωπείται επαρκώς. Δεν είναι εδώ ο εισηγητής οπότε υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν λοιπόν δεν εκπροσωπείται η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στη συζήτηση αυτή αυτό δείχνει μία μια έλλειψη προσοχής σε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Ας δούμε τώρα το θέμα. Δεν νομίζω ότι κανείς ε, είναι ε, ενθουσιασμένος να επιβάλλουμε φορολογία απλώς για να υπάρχει αυτή η επιβολή. Υπάρχει κάποιος λόγος και αυτή τη στιγμή πρέπει να επενδύσουμε διότι έχουμε σημαντικές ανάγκες επενδυτικές που δεν μπορούν να καθυστερήσουν 20 χρόνια και πιστεύω πιστεύω ότι χρειάζεται να επενδύσουμε για να γίνει η ηγετική ευρωπαϊκή οικονομία στον 21ο αιώνα. Και ή θα μειώσουμε το κόστος μας, πράγμα το οποίο είναι ανόητο, δεν θα το πετύχουμε ποτέ, ή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία, να επενδύσουμε στην παιδεία, στην έρευνα, στην καινοτομία και ε, στην υποδομή. Σκεφτείτε πράγματα όπως ε, το European Smart Super για την κατανομή ε, ενεργείας. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί μόνο στο ιδιωτικό τομέας να τα πετύχει, διότι Εάν ε, η περίοδος αποπληρωμής είναι 30 χρόνια, κανείς δεν θα επενδύσει. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε, δεν πρέπει να είναι όμως μόνο δημόσιες επενδύσεις, διότι η ιδιωτική επένδυση των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι, είναι σημαντική, αλλά όχι επαρκής. Πρέπει λοιπόν και να επενδύσουμε και ε, να δαπανίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επιζητήσουμε επιθετικά τις ε, κινήσεις αυτές, να μην μειώσουμε τις επενδύσεις, να έχουμε καινοτόμους πόρους και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας μειώνοντας ε, το, την ε, φορολογία στην απασχόληση και στην εργασία διότι αν θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό εργασίας της ε, δημιουργίας προσθέμενης αξίας θα έπρεπε να ίσως ε, να φορολογήσουμε ε, την ε, ενέργεια αλλά όχι την εργασία. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Οπότε αν συμφωνούμε επί αυτής της αρχής θα πρέπει κάπου να βρούμε τα χρήματα. Όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον αλλά για να βρούμε το τη σωστή πηγή πόρων. Επίσης ε, πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα σε όλα τα δημοσιονομικά θέματα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Δεν υπάρχει 100% αποτελεσματικότητα αλλά στη ζωή μου έχω δει και στον ιδιωτικό τομέα να γίνονται ανόητες κινήσεις να υπάρχει σπατάλη χρημάτων οπότε δεν υπάρχει ιδεατή βελτίστη αποτελεσματικότητα χρήσεως χρημάτων. Λοιπόν, θα πρέπει η Ευρώπη να παίξει έναν ηγετικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια χώρα μόνο δεν μπορεί να το επιτύχει, αλλά μιλάμε για κρίσιμη μάζα. Μία αγορά, αν και μία αγορά δεν καλύπτει τα πάντα, αλλά όταν έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκους μπορούμε ε, να ε, καλύψουμε το ένα στοιχείο και αν ε, κάνουμε ένα απλό σύστημα χωρίς πολλές λεπτομέρειες θα είμαστε αποτελεσματικοί. Θέλουμε λοιπόν κάτι το απλό και αυτό ίσως θα ευχαριστήσει ε, τους ε, Βρετανούς συντηρητικούς ή την, ε, τους φιλελεύθερους αλλά το όλο θέμα είναι το κόστος. Το κόστος αυτής της προσπαθίας είναι αστείο μπροστά στην φορολογία εισοδήματος. Άρα είναι κάτι εύκολο και φθηνό και μ' αρέσουν οι φθηνές λύσεις η ε, φορολόγηση της ενεργείας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η φορολογία πρέπει να καταργηθεί ή ε, να, για να ε, ε, χρηματοδοτήσουμε μία επένδυση που θα γίνει μία φορά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την φορολόγηση της ενεργείας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την υποδομή και να καταργηθεί αυτή η φορολογία, όσο παράλογο και να φαίνεται. Εάν είμαστε καινοτόμοι, πιστεύω ότι ίσως δεν πρέπει να εναρμονίσουμε αλλά να συντονίσουμε ε, την ε, φορολογία των επιχειρήσεων και η CCCB είναι ε, καινοτόμο μέτρο διότι όλοι κακό στον εαυτό μας κάνουμε όσο συντηρούμε αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό. Ε, πρέπει επίσης όπως είπαμε να έχουμε καινοτόμα μέτρα και θα ολοκληρώσω με μερικά γενικά σχόλια. Δεν αναφέρουμε για τον ισοσκελισμό των δημοσίων οικονομικών αλλά ε, εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης διότι αν δείτε τα εκατομμύρια, ε, ε, δισεκατομμύρια που επενδύει η Κίνα αυτή τη στιγμή για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, για τους πυρηνικούς σταθμούς θέλουμε η Ευρώπη να μείνει πίσω, πίσω να γίνει μουσείο ή να ηγεθεί. Εγώ θα προτιμώ προτιμούσα να ηγείται. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι. Και τώρα πηγαίνω σε μία άλλη ιδέα η οποία συχνά συζητείται εδώ που είναι το level playing field αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει level playing field. Εκτός και αν είχαμε παγκόσμια διακυβέρνηση και πιστεύω ότι ούτε τα δυσέγγονά μας δεν θα το δούνε. Δεν θα υπάρξει ένα ενιαίο ισότιμο πεδίο. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε ε, πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης σαν τους Κινέζους. Δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εάν θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια οικονομία κοινωνικής αγοράς, δεν πρέπει να περιμένουμε ο άλλος κόσμος να το πράξει. Εάν θέλουμε να ηγηθούμε ε, τη μετακίνηση ε, του βάρους φορολογίας από την εργασία σε άλλες πηγές, θα πρέπει εμείς να το προτείνουμε. Άρα Θέτω το ερώτημα, οι πολίτες θα πληρώσουν αυτό, είναι πολύ σημαντικό, διότι αναφερόμαστε πρώτον στη δικαιοσύνη, οι πολίτες ούτως ή άλλως πληρώνουν και πληρώνουν ακριβά την ε, οικονομία καζίνου την οποία εφαρμόζουμε. Και όταν λέμε εμείς σαν βουλευτές δεν πληρώνουμε τόσο, Όλοι όμως οι πολίτες πληρώνουν πολλά. Ε, μπορεί λοιπόν να υπάρξει μία πιο δίκαιη αλλά πιο αποτελεσματική ε, φορολογία, δηλαδή δικαιοσύνη της φορολογίας ε, και να χρεώνουμε τις σωστές πηγές και ο, ο δημοσιονομικός τομέας ο οποίος μειώνει την αξία αντί να προσθέτει αξία στην οικονομία είναι ένα μέτρο δικαιοσύνης. Επίσης αποτελεσματικότητα οι πολίτες θα είναι ευτυχείς να πληρώνουν αρκεί να αποδίδει η επένδυσή τους αυτή, να έχουν καλή παιδεία, καλή υποδομή, αποτελεσματική οικονομία. Οπότε με τα χαράς θα πληρώσουν. Οπότε μόνο εάν κάνουμε κάτι τέτοιο θα πάμε μπροστά. Μπορούν αυτό να γίνει βεβαίως αλλά όταν μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να κοιτάμε ότι ε, σωστά επενδύουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι ε, ε, ε, ε, συλλέγουμε και ε, το εισόδημα αυτό σωστά. Επίσης ο Μίχαελ μου θύμισε ότι πρέπει ο καθένας να πληρώνει αυτά τα οποία οφείλει να πληρώνει. Ευχαριστώ. Και θα είμαστε ευτυχείς όταν θα έχουμε κάθε χώρα να παρουσιάζει μία έκθεση. Η Αρλίν. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, διότι νομίζω ότι στο 2011 θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχουμε μια επιτροπή κρίσεως και είναι πολύ σημαντικό η δικιά μας επιτροπή να ηγείται στη διατύπωση των ε, μεθόδων ε, με τις οποίες θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Συμφωνώ με τον Όλε Σμιτ ε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικονομία με τον τρόπο που διατυπώθηκε μας οδήγησε στην κρίση και τώρα ζητάμε από το φορολογούμενο να πληρώσει. Και ε, οι τράπεζες είναι οι μόνες οι οποίες κερδίζουν χρήματα μέσα σε αυτή τη διεργασία τώρα. Οπότε δεν πρόκειται για θέμα έγκλημα και τιμωρία, αλλά πρέπει ο δημοσιονομικός τομέας να αντιμετωπίσει τα λάθη τα οποία έχει κάνει. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μεταρρύθμισης διατυπώσουμε στην Επιτροπή μας και θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ε, φορολογούμενοι ε, πληρώνουν πολύ περισσότερο από ότι π.χ. τα Υπουργεία. Οπότε υπάρχει ανισορροπία και ο στόχος ε, των μέτρων μας είναι να συλλέξουμε περισσότερους πόρους, να υπάρχει μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση του δημοσίου τομέα ή την ανάπτυξη της οικονομίας και να υπάρξει ένα τομέα τομέας διεθνούς ανταγωνισμού χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα λάβουμε το μέτρο να εξασφαλίσουμε ε, πιο υπεύθυνο τομέα δημοσίων οικονομικών. Χαίρομαι διότι η συγγήτηρια δεν κοίταξε μόνο το, τη φορολόγηση της ενεργείας αλλά και τον τομέα της ανάπτυξης και αν είχαμε ε, έναν ε, υπεύθυνο τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν θα χρειαζόταν να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα τώρα διότι ο τομέας αυτός ε, έχει επηρεάσει και τον, της υποανάπτυξης χώρες με ε, την κερδοσκοπία στις πρώτες ύλες. Είναι κάτι το οποίο ίσως δεν έχει εξεταστεί αρχικά γιατί δεν επηρεάζει τόσο την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά περισσότερο τις υποανάπτυξη χώρες. Χαίρομαι ότι ο κύριος Λάμπερτ έθεσε το θέμα των πολιτών διότι οι πολίτες προπορεύονται και ε, ουσιαστικά διπλοπληρώνουν διότι δεν τους ζητάμε μόνο να στηρίξουν τη διάσωση των χρηματοοικονομικών μέσων αλλά ζητάμε να μειωθούν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και δεν πιστεύω ότι οι τράπεζες είναι αμέτωχες σε αυτή τη διαδικασία. Άρα ο πολίτης δεν χρειάζεται να πληρώνει τα διπλά και γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε στις κινήσεις πολιτών οι οποίοι ζητούν επισταμένως να υπάρχει ένας μηχανισμός φορολογίας των χρηματοοικονομικών ε, οργανισμών. Τέλος, ε, νομίζω ότι κάποιος μίλησε για τα κενά. Πρέπει πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν δημόσιες σχέσεις που λέγουν ότι θα ήθελα να υπάρξει μία φορολόγηση των τραπεζών ή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά ρί όπως το Ηνωμένο Βασίλειο να εισπράξουν 2,4 δισεκατομμύρια κριτήρια και τελικά τους ε, επιστρέφουν ένα εκατομμύριο άρα ουσιαστικά δεν τις φορολογούν. Οπότε ε, δεν θα πρέπει από τη μια μεριά να φορολογούμε και από την άλλη να βοηθούμε διότι οι πολίτες δεν είναι βλάκες, ξέρουν ότι ό,τι δίνουμε το ένα χέρι το παίρνουμε από το άλλο και ε, δεν χρειάζεται να ασχολούμε με διαφήμιση και να λέμε ότι είναι υπεύθυνε οι χρηματοοικονομικές οργανώσεις μεν, αλλά εμείς καλύπτουμε τα έξοδά τους από, το από την άλλη πλευρά. Και η δικιά μας επιτροπή πρέπει να είναι πολύ αυστηρή, να διατυπώσει τις εναλλακτικέ λήξεις και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα υπεύθυνα και να κοιτάξουμε ο καθένας να καλύπτει τα δικά του έξοδα, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Υπερβόνσου. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από αυτά τα οποία θα ήθελα να πω τα είπαν ήδη οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Η έκθεση την οποία παρουσίασε η Άννη Ποδηματά είναι κάτι για το οποίο την ευχαριστώ. Είναι τεράστια όμως η έκθεση, η θεματική που καλύπτει. Το θέμα των καινοτόμων χρηματοδοτήσεων καλύπτει τα πάντα, καλύπτει ακόμα και τη φορολογία, γενικά το σύνολο της φορολογίας. Το θέμα το φορολογικό πέραν του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα είναι καινοτόμα, όλα είναι καινούργια. Αν δει κανεί το πώ έχουν εξελιχθεί τα θέματα τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα μένει να γίνουν. Συνεπώ, το έγγραφό σας το λέει αυτό, ότι η καινοτόμος χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο κάποιες επιχειρήσεις, αλλά γενικότερα την δυνατότητα χρηματοδότησης των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση που κάνουμε είναι αναγκαία. Το θέμα του δημοσίου χρέους, το θέμα του ιδιωτικού χρέους καθιστά πολύ δύσκολη και επίπονη την χρηματοδότηση από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην αλλαγή του τρόπου ζωής και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ταυτόχρονα με την γύραση του πληθυσμού. Τεράστιες προκλήσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αυτά από τη μια μέρα στην άλλη ούτε με κάποια κονδύλια και κάποια μετρητά έστω και εξασφαλισμένα. Τίθεται λοιπόν το θέμα σαν ένα ερώτημα εδώ. Σε τι βοηθάει η φορολογία γενικά. Η φορολογία επιτρέπει πρώτον να βρούμε, αν θέλετε, κάποιες μορφές χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες επενδύσεις, τις οποίες θα καλύψει, αν θέλετε, συλλογικά ο πληθυσμός. Ταυτόχρονα όμως η φορολογία είναι και ένα μέσο κοινωνικής ανακατανομής πόρων, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν διαβάζει την έκθεση της ε, κυρίας Ποδήματα. Το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το συζητάμε. Ε, είναι σαν να είναι ταμπού. Το αποφεύγουμε. Στο σύνολο των προτάσεων τις οποίες κάνουμε λοιπόν θα πρέπει να μην ξεχνάμε αυτούς τους δύο στόχους και να προσθέσω και έναν τρίτο στόχο αν μου επιτρέπετε. Να περάσουμε από τη φορολογία της εργασίας σε μια φορολογία στο κεφάλαιο. Αλλά αυτό πάντα άπτεται της ε, κοινωνικής ανακατανομής. Συνεπώς, η χρηματοδότηση, ακόμα και η πιο αποδοτική και η πλέον υποσχόμενη είναι η φορολογία των διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Νομίζω ότι αυτά τα οποία προτείνονται είναι λίγο πιο φιλόδοξα από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Όλε Σμιτ. Γιατί αφορούν το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε τη διεθνή διάσταση, την παγκόσμια διάσταση. Όταν μιλάμε για φορολογία των διεθνών ε, τραπεζικών, πιστοτικών λοιπά ενεργειών και πράξεων, προφανώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε επίπεδο πολιτικής κορυφής οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι γενικά όταν το συζητάνε αυτό συμφωνούν πάνω κάτω και όταν περνάμε στους υπουργούς οικονομικών ή εθνικής οικονομίας όπως θέλετε εκεί υπάρχουν εξαφνικά πάρα πολλές τεχνικές επιφυλάξεις οι οποίες όμως είναι ανυπέρβλητες και οι οποίες ε, τελικά μας οδηγούν στο να πούμε ότι δεν μπορείτε από τη μία να αρνείστε την αύξηση των ιδίων πόρων, να αρνείστε την διεθνή φορολογία αυτών των συναλλαγών. Είναι προφανές ότι εκεί υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα τα οποία πρέπει να κινητοποιηθούν και είναι απαραίτητα για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Πίσω από όλα αυτά για μια ακόμη φορά πρέπει να γίνει η συζήτηση. Η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη, δηλαδή τι θα γίνει με τα χρήματα τα οποία θα συλλέξουμε από τον φόρο αυτό. Το ίδιο που λέγαμε για το φόρο Τόμπιν, σαν παράδειγμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ή θα είναι εσωτερική πόρη για τα κράτη-μέλη, ή θα είναι στην ουσία το κατεξοχήν κυρίαρχο και ευνοούμενο, θα έλεγα, ευνοημένο μέσο χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων. Όχι Αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν και θα πρέπει κάποτε να τα αποφασίσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα η στιγμή. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τον κοινοτικό προπολογισμό σε μια πρώτη φάση και μετά επανερχόμαστε στα υπόλοιπα. Τώρα για την ενέργεια, για τον άνθρακα, για την οικολογία, τον φόρο αυτό όπως θέλετε να τον πούμε. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ γιατί κινητοποιεί ένα μηχανισμό τιμών ο οποίος με τη σειρά του μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για την βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας και καταπολέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Βέβαια, αν διατυπώνουμε με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση, υπάρχει πάντα σε εκκρεμότητα το θέμα της ανακατανομής της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει να το καλύψουμε και αυτό το θέμα, να προσθέσουμε λοιπόν έναν πυλώνα τον οποίο είχα ονοματίσει στην έκθεση Κλίντ στην αρχή, όχι στην τελική βερσιόν, αυτό που είχα ονοματίσει ενεργειακή ασπίδα. Τι είναι αυτή η ενεργειακή ασπίδα. Είναι κάτι το οποίο αν δεν υπάρξει στην ουσία η οικολογική αυτή η φορολογία ή του διεξιδίου του άνθρακα ή του άνθρακα κτλ. θα λειτουργήσει στρεβλωτικά απέναντι στους ασθενέστερους οικονομικά. Γιατί οι ασθενέστεροι οικονομικά είναι αυτοί οι οποίοι θα φυγούν από ε, τον συγκεκριμένο φόρο, ο οποίος επαναλαμβάνω καλύπτει τις κατοικίες ουσιαστικά και καλύπτει τις μεταφορές ουσιαστικά. Οπότε ποιοι φύγονται αυτή η κατηγορία με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Το θέμα των ευρωομολόγων, το θέμα του ευρωπαϊκού δανεισμού είναι καλό που το αναφέρετε γιατί τώρα είναι η στιγμή να το συζητήσουμε, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε το πρώτο βήμα. Έτσι θα χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις τις οποίες έχουμε ανάγκη. Και συμφωνώ επίσης και με τον Φίλιπ Λάμπερτ στην ιδέα που έχει σχετικά με την εναρμόνιση των φορολογικών βάσεων. Ε, είναι και εδώ θέμα, αν θέλετε, φορολογική καινοτομίας. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε ε, να το κρύψει στα ντουλάπια της το θέμα αυτό στην αρχή της ε, εντολής της. Τώρα έχει αρχίσει και έρχεται στην επικαιρότητα πάλι. Και υπάρχει επίσης το θέμα και της φορολόγησης ε, της αποταμίευσης. Και εδώ υπάρχουν καινοτόμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν όπως το ότι τα τράστα ας πούμε θα πρέπει να υποστούν τέτοιου είδους φορολογικές παρεμβάσεις και υπάρχουν πολλά στοιχεία στην ε, έκθεση αυτή εργασία, στο κείμενο εργασίας και θα πρέπει ίσως να προσθεθούν και άλλα. Και άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Να δούμε πώς θα προσπαθούμε. Δεν ξέρω, δεν γίνεται να μιλήσουν όλοι. Ο πρώτο. πρώτος. Και αν άλλος δεν ζητήσει το λόγο, προσπαθήσουμε τους όλοι. Αλλά πρέπει και η Επιτροπή να λάβει το λόγο για να μας πει τι έγινε όσον αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων, ε, ε, αν γίνεται. Ναι. Μετά από όσα έχουν λεχθεί μπορώ να περιοριστώ σε λίγα μόνο σημεία. Δηλαδή αν ισχύουν τα στοιχεία που έχω τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά διαθέτει 20-30% ε, του ΑΕΠ των χωρών ε, για την προστασία των τραπεζών και εδώ δεν αναφέρομαι ε, εις τον κρατικό προϋπολογισμό δηλαδή εάν τα στοιχεία αυτά είναι σωστά αντιπροσωπεύουν 16% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο Σχετικά, κοιτάζοντας λοιπόν αυτούς τους αριθμούς, ο συνάδελφος Στέλτσεκ δεν είναι εδώ πια, αλλά δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά το ουσιαστικό ερώτημα είναι πόσο καιρό θα θα αντέξουν οι φορολογούμενοι να χρηματοδοτούν την κρίση αυτή. Ή την επόμενη, αυτό θα είναι το επόμενο ερώτημα η οποία θα προκύψει και όταν πηγαίνουμε στις εκλογικές περιφέρειες ε, με συναδέλφους ε, πρέπει να εξηγήσουμε διάφορα θέματα. Παραδείγματο χάρη, σήμερα το πρωί αγοράσατε ένα εργασιών για οτιδήποτε έχετε καταναλώσει. Και γιατί αυτή ή ένα ποτήρι τσάι ή έναν καφέ ή το μεσημέρι στην καντίνα γιατί θα πληρώσετε το φόρο ε, κύκλου εργασιών ε, για, για οτιδήποτε έχετε καταναλώσει και γιατί αυτοί οι οποίοι αυτό αυτόματα κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ μέσω αγοραπολισιών και κινούνται αυτοματοποιημένα δεν πληρώνουν φόρο κύκλου εργασιών. Ε, πηγαίνετε στην, σε οποιαδήποτε εκλογική ε, περιφέρεια και δέστε τι λέει ο κόσμος. Γιατί πρέπει να πληρώσει κανείς το φόρο κύκλου εργασιών για ένα καφέ ή για ένα τσάι και γιατί ε, ε, στέλνουμε στις αποχετεύσεις κατευθείαν τα δισεκατομμύρια ε, των τραπεζικών συναλλαγών και κάποια στιγμή θα πρέπει να χρειαστεί να, να γίνει αυτή η συζήτηση ποιος θα χρηματοδοτήσει την επόμενη κρίση πού θα βρεθούν τα χρήματα και γιατί δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ο συνάδελφος Λάμπερς είπε ποιος θα ηγηθεί. Εντάξει. Να, να ηγηθούμε, αλλά θα σου πω κύριε Λάμπερτ τι θα γίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι το Συμβούλιο ε, θα πηγαίνει σε μία διεθνή συνάντηση, θα γυρίσουν και θα μας πούνε ο καιρός είναι κακός, οι άλλοι δεν μας βοηθάνε, τα πράγματα είναι δύσκολα, είμαστε σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί, ε, χρειάζεται να γίνει ακόμη ε, μία μελέτη να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση αν δεν κάνουμε τίποτα Τέτοιε τέτοιες συζητήσεις θα κάνουμε και ε, λυπούμε. Εγώ δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να κάνω τέτοιες συζητήσεις και πιστεύω ότι η, Επιτροπή αυτή πρέπει να σέβεται την εργασία που κάνει, να μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες για τη δουλειά που κάνει και θα έπρεπε να πούμε σε όλους, όχι μόνο στη δικιά μου πολιτική ομάδα, αλλά σε όλους, ότι όχι κύριοι, αυτό πλέον δεν μας ικανοποιεί και η εντολή μας έχουν δώσει οι πολίτες ε, μας λένε κάτι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να πληρώνει. Είναι θέμα εξυπνάδας. Πρέπει όμως να έχουμε το θάρρος να απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο τίθεται. Θα χρειαστούμε την σύμπραξη όλων των πολιτικών ομάδων ε, του Κοινοβουλίου αλλά δεν είναι μόνο θέμα των συντονιστών. Καλό είναι να ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρονται και ποιοι όχι. Σας παρακαλώ όλοι πρέπει να συνεργαστείτε επικοδομητικά για να μπορέσει να επιτύχει εδώ το Κοινοβούλιο διότι αυτό ζητάει από εμάς οι πολίτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί είναι εξαιρετική και πυκνή η κατεύθυνση που έδωσε στη συζήτησή μας η κυρία Ποδηματά και ταυτόχρονα πολλά από αυτά τα οποία ήθελα να πω ακούστηκαν από τους συναδέλφους. Δεύτερο, ένα ερώτημα πολιτικού τύπου, το οποίο συνδέεται αν θέλετε με την ε, εξαιρετική παρουσίαση την οποία έκανε ο Μπούλμαν. Στις 12 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, εμείς έχουμε τη συνάντηση ε, στη Σεούλ της ομάδας των 20, του G20. Διαρωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πάρουν μέρος στη συνάντηση της Σεούλ, με τι εντολή θα πάνε εκεί για να συζητήσουν αυτά τα οποία λέμε τώρα δηλαδή για την καινοτόμο χρηματοδότηση, όπως επίσης και για τη φορολογία των τραπεζικών και γενικότερα συναλλαγών αυτών. Συνεπώς, από ό,τι φαίνεται, στο θέμα της φορολογίας των, των ε, τραπεζικών συναλλαγών, ουσιαστικά όλοι κρύβονται. Κρύβονται ο καθένας πίσω από ένα άλοθη. Εμείς ναι μεν συμφωνούμε, αλλά τελικά οι υπόλοιποι δεν συμφωνούν, λέει ο ένας. Το θέμα είναι, λένε ορισμένοι, ότι για να κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε μόνο σφαιρικά. Συνεπώς τίθεται εδώ το ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό κόκκινο βούλιο. η δική μας Επιτροπή, επί τη βάση της συζήτησης την οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα εδώ και 1,5 χρόνο και με τις προτάσεις τις οποίες κάνει η κυρία Ποδηματά μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις μας πριν από τη συνάντηση των 20 έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική προσπάθεια της Ευρώπης όπως είπε ο Ούντο να επιδιώξει τους στόχους της καινοτόμου χρηματοδότησης και της φορολογίας αυτών των συναλλαγών σε σφαιρικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας προσπαθήσουμε αυτό τουλάχιστον να κάνουμε. Τελειώνω. Υπάρχει κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Ούντο και το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Μας ενδιαφέρει όλους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αγορές είναι πολύ πιο γρήγορες από εμάς. Συνεπώς, τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε εμείς σε φαινόμενα τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σήμερα ότι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, όπως το light frequency trading. Στις χρηματαγορές υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τρόπο θα έλεγα διάθεσης επιβολής κυρώσεων, αλλά θα πρέπει να επιτρέψουμε στις ίδιες τις αγορές να λειτουργήσουν καλύτερα από ό,τι λειτουργούν σήμερα. Ε, ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πρόκειται για μια έκθεση πάρα πολύ εύστοχη και επίκαιρη. Και έχουμε τρεις λόγους ε, για αυτό. Πρώτα-πρώτα, η οικονομική διακυβέρνηση Δεύτερον, κρίση. Και τρίτον, η αναγκαιότητα για μια ανοιχτή και παγκόσμια οικονομία όσον αφορά την κρίση. Νομίζω ότι το ουσιαστικό είναι ότι η κρίση μας έδειξε ότι για μία μεγάλη περίοδο κάποιοι λίγοι κερδίζανε και τελικά όλοι πλήρωσαν την ύφη. Για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση χρειάζεται να υπάρξει εποπτική δράση κανονιστική, ρυθμιστική δράση αλλά και διορθωτική φορολογική παρέμβαση. Είναι συστημικό αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, συστημικής φύσης για εγγυήσεις δηλαδή, ε, για ε, θωράκιση, για πλαισίωση του συστήματος και έτσι να ε, αντιδράσουμε για την κρίση. Δεύτερον, από πλευρά διακυβέρνηση. Το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε ένα πλέγμα κανόνων. διακυβέρνηση θα πει σίγουρα κανόνε, αλλά σημαίνει επίση και αρχέ, στόχου μέσα. Και ξέρουμε ότι μιλούμε για μέσα, μια που σήμερα η Ευρώπη περισσότερο από πότε διαπιστώνει πόσο το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ και οι δαπάνες πρέπει να συγκρατηθούν. Είδαμε τι έγινε με τα ευρωομόλογα, είδαμε τι γίνεται στην εσωτερική αγορά και ότι επομένως θα πρέπει να συνεχίσουμε να αριστοποιούμε τις φορολογικές αποδόσεις. Άρα χρειάζεται μια τέτοια παρέμβαση. Τρίτον, θα πρέπει να μπορέσουμε το φορολογικό σύστημα να προσαρμοστεί σε μια ανοιχτή οικονομία. Χρειάζονται επομένως σημαντικές αλλαχές να προσαρμοστούμε σε ένα καινούριο σύστημα όπου θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε αυτό το τέλος στις ε, συναλλαγές αλλά να μην τις επιβαρύνουμε δύο φορές γιατί υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία δεν θα πρέπει να φορολογηθούν και μάλιστα με τρόπο έμεσο. Αν θέλουμε παγκόσμια και ανοιχτή οικονομία, τότε θα πρέπει να παράσχουμε εγγύσει ότι δεν πρόκειται να ανέβει κι άλλο το, το κόστος της δαπάνη, η δαπάνη ε, το κόστος τη εργασία. Και επίσης να κάνουμε κάποιε διορθωτικέ κινήσεις όπου το σύστημα δεν είναι σταθερό και όπου το φορολογικό σύστημα τη χρειάζεται κοινέ προσπάθειε να δούμε οπωσδήποτε πώς θα βρούμε νέους πόρους, αλλά τελικά το ερώτημα το οποίο εκρεμεί είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση. Έχουν πολλά αλλάξει και άρα χρειάζεται ένα νέο σύστημα δημοσιονομικό το οποίο να αντιστοιχεί στις νέες συνθήκες. Στην οικονομία που πραγματικά σήμερα υπάρχει. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, όπως σας προείπα έχουμε εκπροσώπους της Επιτροπής και τον Μάρτιο ε, είχαμε αυτό το ψήφισμα, το Μάρτιο ζητήσαμε ε, μελέτη επιπτώσεων. Παρακαλώ. Πέστε μας, αλλά αφήστε λίγο χρόνο τόσο να μπορεί κύριε Ποδηματά να απαντήσει σε αυτά τα οποία ε, ακούσαμε ήταν τόσο ενδιαφέροντα. Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας τονίσω ότι ασχολούμεθα εντατικά στην Επιτροπή με το θέμα αυτών των νέων ε, μέσων χρηματοδότησης και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Είπαμε ότι θα υπάρξει ε, μια ανακοίνωση όσον αφορά αυτήν την ε, φορολόγηση των συναλλαγών. Και θα σας ενημερώσουμε. Άνι, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Σάρων. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδους συζητητές όσους πήγαν το λόγο ε, γιατί θεωρώ εξαιρετικά επικοδομητική την συζήτηση που έγινε και τις προτάσεις που ακούστηκαν. Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα ζήτημα που προκαλεί ε, διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχουν διαφορετικές ε, γνώμες. Είμαστε στην αρχή της συζήτησης και θέλω να πιστεύω ότι χτίζοντας πάνω ε, στην κοινή βάση, διότι υπάρχει μια κοινή βάση και νομίζω ότι το ανέφερα και εγώ στην εισαγωγική μου παρέμβαση, αλλά και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους, η συζήτηση δηλαδή που κάνουμε σήμερα γύρω από τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και την αναζήτηση νέων πόρων, ε, χρηματοδότησης μεγάλων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων στόχων, νομίζω ότι αναγνωρίζεται από τους ε, περισσότερους ότι συνδέεται ε, με τη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται για την οικονομική διακυβέρνηση και με την προσπάθεια που γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να θεσπίσουμε καλύτερους και αποτελεσματικότερους κανόνες εποπτείας και λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη ε, αφορά στο εξής. Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε φορά ε, που ανοίγει συζήτηση για ζητήματα φορολογίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο διατυπώνονται εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις. Στην πραγματικότητα όμως μπορούμε να κουβενιάζουμε σήμερα για τον στενότερο οικονομικό συντονισμό, για την εγκαθίδρυση μιας οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, χωρίς να ακουμπάμε στα ζητήματα της φορολογίας, Υπάρχει εκεί εξαντικειμένου νομίζω ένα πολύ μεγάλο νοητικό κενό ε, το οποίο θα πρέπει να το ε, υπερβούμε, να το συγκαλύψουμε. Είναι η στιγμή που θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να προωθούμε τα ζητήματα της εναρμόνισης αλλά και να μιλάμε για ευρωπαϊκούς φόρους, έσοδα δηλαδή, που θα μας επιτρέψουν σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, σε μια συγκυρία όπου η κρίση βρίσκεται ε, ακόμα σε εξέλιξη, οι εθνικοί προπολογισμοί στα περισσότερα κράτη-μέλη συμπιέζονται, υπάρχουν περικοπές, ουδή συζητάει σοβαρά ε, την αύξηση των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα κράτος μέλος στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται ε, για τον προϋπολογισμό και για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν συζητάει την αύξηση της συμβολής του στον κοινοτικό προϋπολογισμό και ταυτοχρόνως έχουμε μπροστά μας πολύ φιλόδοξα σχέδια Ορισμένα από αυτά περιγράφονται στη στρατηγική 2020. Υπάρχει η χρηματοδότηση των στόχων της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής που αποτυπώνονται στο πακέτο της ενέργειας και του κλίματος που ψηφίσαμε πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει η προσπάθεια για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ως εκ τούτου δημιουργείται ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς ε, όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια θα χρηματοδοτηθούν. Εκεί λοιπόν έρχεται η συζήτηση για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία να καλύψει ένα κενό. Δεν είναι μόνο εκεί που θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Και όπως είπαν αρκετοί συνάδελφοι, δεν είναι μόνο τα ζητήματα που αφορούν στη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχουμε στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας να μιλήσουμε για τα ευρωομόλογα. Δεν το έφερα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, ένα σημαντικό θέμα που έχει έρθει στο προσκήνιο και χρήζει ε, απαντήσεων, ε, καινοτόμα λοιπόν χρηματοδοτικό εργαλεία με την έννοια των μη παραδοσιακών. Δεν βρίσκω να υπάρχει τίποτα το περίεργο και πολύ, περισσότερο τίποτα το ύποπτο ε, στον όρο καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα, νέοι φόροι. Δεν μιλάμε στην πραγματικότητα για νέους φόρους με την έννοια ότι αυτό βασικό ζητούμενο σήμερα είναι ε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να συμβάλλουν κατά το δυνατόν με δικαιότερο τρόπο στα φορολογικά έσοδα όλοι εκείνοι οι οποίοι μέχρι σήμερα εξαιρούνται από τα φορολογικά βάρη. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, έχουν το μεγάλο μερίδιο του βάρους αυτή τη στιγμή, το επομίζονται αυτοί. Ε, ο χρηματοπιστωτικός τομέας χωρίς καμία διάθεση εκδίκησης και τιμωρίας ε, ε, αυτά όλα μακριά από εμάς. Συνυπολογίζοντας όμως το γεγονός ότι τα, την τελευταία δεκαετία με βάση όλες τις έρευνες που έχουν ε, δημοσιοποιηθεί, το τελευταίο διάστημα ο όγκος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κάθε είδους εκτοξεύτηκε στα ύψη έφτασε να είναι το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Υπήρξε, αντικατοπτρίστηκε αυτή η τεράστια αύξηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με κάποιο τρόπο στην ανάπτυξη της ε, παγκόσμιας οικονομίας. Λέω λοιπόν ότι ε, το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε νέα φορολογικά βάρη σε αυτούς που επομίζονται ήδη σημαντικά φορολογικά βάρη, πολύ περισσότερο στη σημερινή συγκυρία. Το θέμα είναι ε, εφόσον αναγνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ανάγκη από καινούργια έσοδα, να βρούμε τρόπους ώστε ε, τα έσοδα αυτά να τα συγκεντρώσουμε με έναν δικαιότερο τρόπο από ό,τι τα συγκεντρώνουμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευτυχώς υπήρξε ο χρόνος. Προθεσμία λοιπόν προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου, 12 Νοεμβρίου οι τροπολογίες, συζήτηση στις 30 Νοεμβρίου, επανεξέταση τροπολογιών στις 24 Ιανουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 25 Ιανουαρίου, Ολομέλεια 2η του Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες τις οποίες θα επεξεργαστεί και θα μας καταθέσει εκ νέου. Θα τα πούμε το απόγευμα ελπίζω.